Kolleginnen und Αγαπητοί συνάδελφοι, Σας έχουμε στείλει ηλεκτρονικά τη νέα ημερήσια διάταξη. Ηλεκτρονικά δεν είναι ακόμα διαθέσιμη. Έχουν γίνει κάποιες αλλαγές. Έχουμε 5.30 με 6.30 το απόγευμα μια ανταλλαγή απόψεων σε σχέση με τις κατηγορίες οι οποίες έχουν διατυπωθεί σε σχέση με την EULEX, την EULEX στο Κωσυχοπαίδιο. Και θα συζητήσουμε εδώ με, την, ε, με τον κύριο Κένεθ ο οποίος είναι επικεφαλής της ε, υπηρεσίας ε, μη στρατιωτικών υποθέσεων και τον Φερνάντο Τζεντιλίνη, ο οποίος είναι διευθυντής για την ε, Δυτική Ευρώπη και τα Βαλκάνια της υπηρεσία Εξωτερικών, ε, Εξωτερικής Επομένω, Επομένως, εδώ είναι θέμα του ελεγκτικού ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα πρέπει να εξετάσουμε τα θέματα αυτά. Υπάρχει κάποια αντίρρηση σε σχέση με τη μερική διάταξη ανακοινώσει του Προέδρου. Έχουμε τον κύριο Πλένκοβιτς αύριο, από ό,τι γνωρίζω. Μάλλον την εκλογή του κύριου Πλένκοβιτς και θα έχουμε συζήτηση με την ε, συζήτηση για τα γεγονότα στην Ουκρανία και συγκεκριμένα τις παράνομες εκλογές στο Λούγκανς και στο Ντόνετσκ. Θα πρέπει να συζητήσουμε αυτά τα θέματα με την ε, αρμόδια για τα θέματα αυτά, επικεφαλής της Επιτροπής ε, Παρακολούθησης. Για τα πρακτικά, αν έχετε αντιρρήσεις, δεν έχετε αντιρρήσεις, μπορούν να θεωρηθούν ότι έχουν εγκριθεί λοιπόν και τα πρακτικά και ερχόμαστε τώρα στο Νότιο Κάφκασο και τις ε, πολεμικές ενέργειες στην ε, Γεωργία. Ο κύριος Herbert Σάλμπερ είναι ο ειδικό εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Νότιο Κάφκασο και ευγενώς έχει έλθει να μας παρουσιάσει τα στοιχεία σε σχέση με την περιοχή αυτή και να προβεί σε μια ανταλλαγή απόψεων μαζί μας και να μας παρουσιάσει λοιπόν την έκθεση που έχει προετοιμάσει για τα θέματα αυτά και είναι έτοιμος επίσης να συζητήσει και τα άλλα θέματα τα οποία μπορεί να σας φανούν ενδιαφέροντα. Και φυσικά και ο εισηγητής της Επιτροπής μας μπορεί να λάβει το λόγο για τα θέματα αυτά. Θα αφιστώ τις απαραίτητες παρουσίες και θα δώσω μέσα το λόγο στον κύριο Σάιμπερ. <coughs> σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ και καλημέρα σας κύριε και κύριοι to brief you on the situation in the South Caucasus and in my on my efforts to implement the mandate that was given to me from 1st of July onwards as EU Special Representative on... Μα το είναι πατημένο αριστερά το κουμπί και δεν φεύγει, δεν πηγαίνει. What did I do so far in the first months of my mandate? Τους πρώτους μήνες, τους πρώτους μήνες της θητείας μου διαχειρίστηκα δύο γύρους των διεθνών διαπραγματεύσεων για τη Γεωργία στη Γενέβη και χρειάστηκαν και πολλές μετακινήσεις στην περιοχή για να μπορέσω να γνωρίσω όλους τους παράγοντες και δυνάμεις στην περιοχή εκεί, καθώς και τις δικές μας δυνάμεις, όπως και εκείνους που θέλουν να αποσχιστούν και εγώ και η υπηρεσία μου μπορέσαμε να τους συναντήσουμε αντίθετα από άλλους διεθνείς παράγοντες που αντιμετώπισαν περισσότερους περιορισμούς. Θα ήθελα να τονίσω το διεθνή χαρακτήρα της εντολής μου που καλύπτει όλο τον Νότιο Κάυκασο και όπως σας είπα, το σημαντικό είναι ότι είχαμε πρόσβαση και στις μη αναγνωρισμένες οντότητες. Προσπάθησα να συνεργαστώ όσο το δυνατόν περισσότερο και με τις άλλες, ε, τους εκπροσώπους των υπολείπων χωρών μελών εκεί, δηλαδή αντιπροσωπιών, στο Μπακού, στο Γερεβάν, αλλά και στη Γεωργία. Η εντολή γενικότερα έχει τρία συστατικά. Το πρώτον, αυτό που σας είπα ίδια επαφές στη Γενέβη, τη διεθνεί διαπραγματεύσει δηλαδή για τη Γεωργία, μαζί με τον ΟΗΕ, τον ΟΗΕ και τον ΟΣΑ, ΟΑΣΕ. Και εγώ έπαιζα το ρόλο πρίμους inter pares σε αυτές τις διαδικασίες. Γενικότερα σχετιζόμενες με τη διαχείριση και λύση της διαμάχης στη Γεωργία καθώς και την εφαρμογή της πολιτικής της Ένωσης ως προς την μη αναγνώριση των αποσχιστικών οντοτήτων. Και το τρίτο συστατικό ήταν η κατάσταση στον Αγκόρνο Καραμπάχ. Πριν αναφερθώ στα τρία αυτά στοιχεία θα θέλω να πω κάτι γενικότερο. Όπως φαντάζεστε η κατάσταση στην Ουκρανία έχει επιπτώσεις και σε αυτά που κάνουμε εμείς εκεί γιατί επηρεάζει πολύ την οτροπία των συνομιλητών μας. Στο Αζερβαϊτζάν ας πούμε η κυβέρνηση με βάση αυτά που γίνονται στην Ουκρανία επιμένει περισσότερο ως προς τη, το ρόλο που παίζει η Ένωση για την εδαφική ακαιρεότητα. Στη Γεωργία η κυβέρνηση θεωρεί στα γεγονότα, βλέπει στα γεγονότα της Ουκρανίας μία επιβεβαίωση και επανάληψη αυτών που έγιναν στη Γεωργία. Προηγουμένως θα θυμάστε εκείνον τον πόλεμο και Όλα αυτά επικρέμανται λοιπόν σαν νέφος από πάνω μας εκεί στο νότιο Κάυκασο. Τώρα μερικά λόγια για το κύριο μου θα έλεγα θέμα της διεθνή συζητήσεις στη Γενέβη που έχουν γίνει από το 8, από τότε που άρχισε η διαμάχη. Εγώ είχα την ευχαρίστηση να συμμετάσχω στον 21ο γύρο που έγινε τον περασμένο Ιούνιο. Εν τω μεταξύ τον Οκτώβριο έγινε κι άλλος ένας γύρος και οδηγούμαστε τώρα προς τον 30ο τον Δεκέμβριο. Ίσως να θυμάστε ότι από την αρχή των διεθνών αυτών συζητήσεων της Γενέβης αναμενόταν να τελειώσουν σε ένα-δύο χρόνια, να είχαν λυθεί όλα τα προβλήματα αλλά είδαμε ότι δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Ακόμα συνεχίζεται ο διάλογος και φτάνουμε στον 300 πλέον γύρο. Από αυτό μπορείτε να καταλάβετε ότι η δυνατότητα να λυθούν ή και να συζητηθούν απλώς σοβαρά αυτά τα προβλήματα είναι κάτι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί. Δεν μπορούν εύκολα οι δύο πλευρές να κάνουν υποχωρήσεις γιατί οτιδήποτε συζητιέται εκεί πολιτικοποιείται αμέσως και αν και οι ίδιες οι συζητήσεις στη Γενέβη δεν αφορούν θέματα καθεστωτικά και οι δύο ή μάλλον όλες οι πλευρές τα βλέπουν όλα υπό το πρίσμα του πώς επηρεάζει αυτό το καθεστώς μου ή και το γόητρό μου ακόμα. Όποτε λοιπόν συζητάμε κάποιο από αυτά τα θέματα, πάντα χρωματίζεται από αυτό το παράγοντα, χρωματίζονται. Έτσι αντιμετωπίζουμε τη δυσκολία ότι στη Γενέβη γενικά είναι οι συζητήσεις πολύ ευπαθείς ε, σε πολλές περιπτώσεις. Δεν μπορέσαμε να συζητη... μπορούσαν να συζητηθούν τα θέματα όπως έπρεπε, αλλά απειλούσαν οι διάφορες πλευρές να αποχωρήσουν αν κάποιο θέμα που τους ενδιέφερε ιδιαίτερα δεν συζητιούνταν όπως ήθελαν εκείνοι. Αυτό έγινε και την πρώτη φορά που πήγα τον Ιούνιο έγινε μια διαμάχη για ένα θέμα της ημερήσιας διάταξης γιατί οι Αμπχάζοι αρνήθηκαν να το συζητήσουν και ήθελαν να αφαιρεθεί τελείως από την ημερήσια διάταξη ενώ οι Γεωργιανοί διαφωνούσαν με αυτό κτλ. Οι Οσετιανοί και οι Αμπχάζοι λοιπόν απεχώρησαν και δεν μπόρεσε να συζητηθεί καθόλου. Τον Οκτώβριο τα πράγματα πήγαν πολύ καλύτερα, συζητήσαμε, μπορέσαμε να συζητήσουμε όλα τα θέματα και σημειώθηκαν και μερικά ανοίγματα από μερικές πλευρές ώστε μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι διεθνείς συζητήσεις της Γενέβης μπορούν να οδηγήσουν κάπου σε κάποιο αποτέλεσμα. Γι' αυτό όμως θα απαιτούνταν ε, περισσότερες και μακρύτερες συζητήσεις που ελπίζω να γίνουν. Από ό,τι σας είπα ίσως βλέπετε ήδη ότι η Γενέβη δεν είναι μέρος όπου μπορούμε να αναμείνουμε επιλύσεις πολλών σειράξεων ή διαμαχών γιατί οι ενδιαφερόμενοι τη χρησιμοποιούν τις συζητήσεις ως μάλλον εργαλείο για αποφυγή περαιτέρω διαμαχών και σειράξεων αλλά όχι για επίλυση υπαρχουσών. Η επιτόπου κατάσταση πολιτική ιδίω, είναι αρκετά τεταμένη. Υπάρχουν ακόμη εντάσεις επιτόπου και γι' αυτό καλό είναι να υπάρχει αυτό το βήμα και όταν λέω στους ενδιαφερόμενους, τους συμμετέχοντες, όταν τους ρωτάω αφού χρειάζεστε αυτό το βήμα γιατί το θέτετε σε κίνδυνο, τότε όλοι λένε ναι το θέλουμε, είναι απαραίτητο Υπάρχουν πολλά θέματα που πρέπει να συζητηθούν και ελπίζουμε και εμείς να καταλήξουμε σε συμπεράσματα, αλλά υπάρχει η επιτόπου κατάσταση που καθιστά αδύνατη κάθε πρόοδο. Τελικά ελπίζω παρόλα αυτά να μπορέσουν να γίνουν, να πραγματοποιηθούν ορισμένοι γύροι επικοδομητικά για να μπορέσουμε να κάνουμε και εμείς κάποια πρόοδο. Κάποιες επιπλέον παρατηρήσεις τώρα για τις προσπάθειες επίλυσης γενικότερα των προβλημάτων στη γεωργία, του προβλήματος της γεωργίας. Εμείς εδώ σαν Ευρωπαϊκή Ένωση και σαν αντιπροσωπεία προσπαθούμε να προχωρήσουμε σύμφωνα με τις γραμμές και τους στόχους που έχει θέσει η Ένωση. Από τη μία, μία αναγνώριση των οντοτήτων που έχουν αποχωρήσει, από την άλλη όμως προσπάθεια επαφών μαζί τους. Είναι ανοιχτό το γραφείο, το δικό μας, ιδιαίτερα προς την πλευρά της Αμπχαζίας. Προσπαθούμε να έχουμε διάλογο με τους κατοίκους της Αμπχαζίας, να δείξουμε ότι είμαστε παρόντες και είναι πιο δύσκολα τα πράγματα με την Νότια Οσετία βέβαια γιατί δεν είναι τόσο επικοδομητική η Νότια Οσετία όσο είναι η Αμπχαζία. Πάντως και με αυτούς προσπαθούμε να έχουμε ανοιχτή πόρτα. Ε, διευκρινίσαμε στην κυβέρνηση της Γεωργίας ότι οι επαφές αυτές που έχουμε είναι προς όφελός τους, διότι τελικά αυτό που θέλει η κυβέρνηση της Γεωργίας είναι οι οντότητες αυτές οι εθνικές να επιστρέψουν στη δημοκρατία της Γεωργίας. Ως εκ τούτου πρέπει να προσπαθήσουμε να εργαστούμε μαζί τους, να τους επηρεάσουμε, να προσπαθήσουμε να επηρεάσουμε τις συνειδήσεις αν θέλετε ε, και τις νοοτροπίες έτσι ώστε σεβόμενοι τις διαφορές να υπάρξει μια ενότητα της χώρας ε, να επιστρέψουμε σε αυτά τα οποία κάποτε υπήρχαν στην Γεωργία, να συνεχιστεί ο διάλογος και να αναπτυχθεί αν είναι δυνατόν ακόμα περισσότερο. Αυτό σημαίνει ότι προσπαθούμε να είμαστε δραστηροί και στα πλαίσια της εφαρμογής μέτρων εμπιστοσύνης, της επαφής και του κοινού εδάφους ανάμεσα στις διαφορετικές εθνικές οντότητες. Προσπαθούμε επίσης να παρακολουθούμε από κοντά την κατάσταση στη Γεωργία. Ε, βλέπουμε ότι η κατάσταση θα μπορούσε να χειροτερεύσει στο μέλλον, ιδιαίτερα το θέμα των μειονοτήτων όπως των Αρμενίων που κατοικούν στο νότιο τμήμα της χώρας, της Γεωργίας, και ε, είναι σε επαφή φυσικά ε, με την κυβέρνηση της Γεωργίας. Τώρα για το Άνω Καραμπάχ. Από την αρχή προσπαθήσαμε να έχουμε καλές σχέσεις με την ηγεσία και στο Γερεβάν και στον Μπακού αλλά και με τους συμμετέχοντες ε, στην ομάδα του Μίνσκ. Οι θέσεις της Ένωσης είναι σαφείς. Εμείς στηρίζουμε τους στόχους της ομάδας του Μίνσκ για επίλυση του προβλήματος. Η διπλωματία σε επίπεδο κορυφής έχει ξαναρχίσει με την συνάντηση κορυφής στο Σότσι τον Αύγουστο, ε, το Σεπτέμβριο και εδώ και μία εβδομάδα στο Παρίσι μετά από πρόσκληση του Γάλλου Προέδρου της Δημοκρατίας. Σαν Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρουμε, είμαστε στη διάθεση ε, των ε, εμπλεκομένων για να κάνουμε προτάσεις για νέα μέτρα εμπιστοσύνης, για συνάντηση και επικοινωνία των κοινοτήτων από την Αρμενία, το Άνω Καραμπάχ και το Αζερβαϊτζάν, έτσι ώστε να υπάρχει ένα επίπεδο αμοιβαίας κατανόησης και να μπορέσουμε από κάποια στιγμή και μετά να εργαστούμε σε πιο συγκεκριμένη βάση. Το να κάνει κανείς προσπάθεια στον τομέα των μέτρων εμπιστοσύνης σε αυτήν την περιοχή του Καυκάσου είναι δύσκολο γιατί οι πλευρές απορρίπτουν με τον έναν τρόπο ή τον άλλο τις συγκεκριμένες αυτές προτάσεις. Η πολιτική ένταση είναι πάρα πολύ υψηλή και αυτό οδήγησε και σε θύματα. Υπήρξαν 50 θύματα στην διαχωριστική γραμμή, πολύ περισσότερα δηλαδή από ό,τι τον προηγούμενο χρόνο. Το Άνω Καραμπάχ λοιπόν δεν είναι ένα μια παγωμένη σύγκρουση θα λέγαμε, είναι μια σύγκρουση εν θερμό και η οποία μπορεί να δώσει κλιμάκωση ε, πάρα πολύ σύντομα. Προσπαθούμε να κατανοήσουμε λοιπόν την κατάσταση και των εκτοπισμένων πληθυσμών από τις συγκρούσεις των τελευταίων 25 χρόνων. Στον Πακού πρόσφατα επισκέφθηκα κάποιες κατοικίες και καταβλισμούς εκτοπισμένων κατάλαβα το τι κάνει η κυβέρνηση των Αζέρων από τη μία και από την άλλη όμως διαπίστωσα ότι οι συνθήκες διαβίωσης ε, είναι πραγματικά ανυπόφορες. Ελπίζω λοιπόν ότι σχετικά με τη σύγκρουση αυτή μια λύση δεν είναι κάτι το οποίο δεν συζητιέται. Είχαμε επαφή με τους συμπροέδρους της ομάδας του Μίνσκ στην τελευταία συνάντηση στο Παρίσι και ο πρέσβης Βόλικ των Ηνωμένων Πολιτειών είναι αισιόδοξο ότι τα πράγματα ακολουθούν μια καλή κατεύθυνση, αλλά ταυτόχρονα δεν έχουμε και ψευδεστήσεις, γιατί στο τέλος η θέση της Μόσχας, η θέση της ρωσικής ηγεσία θα είναι το καθοριστικό στοιχείο για την πιθανή επίλυση μιας λύσης ή όχι. Ε, συνάντησα με την, ηγε... ηγεσία επίσης και στον Πακού και στο Γερεβάν ζήτησα να έχω ελεύθερη πρόσβαση στο Άνω Καραμπάχ να συμφωνούν στις μετακινήσεις μου εκεί έτσι ώστε να μπορώ ε, άμεσα εγώ ίδιος να διαπιστώνω την κατάσταση και να βλέπω ποιες είναι οι προσδοκίες ε, των κατοίκων του Ναμπγκόρνο Καραμπάχ. Ε, αυτό είναι δύσκολο γιατί οι Αζέροι προς το παρόν δεν δείχνουν να επιτρέπουν μια τέτοια δυνατότητα για το Άνω Καραμπά. Αλλά πάντως διευκρίνησα προς τον πρόεδρο του Αζερβαϊτζάν και το Υπουργό Εξωτερικών ότι θα, επιγίνω, ε, θα επιμείνω προς την κατεύθυνση αυτή. Κλείνω εδώ. Είμαι στη διάθεσή σας για πιθανές ερωτήσεις και παρατηρήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Το κύριε Στέτινερ. Σας ευχαριστώ μου δίνετε το λόγο κύριε Πρόεδρε. Κύριε Ζάιμπα, συγχαρητήρια για το διορισμό σας σε αυτή την ευραλική θέση. Χαίρομαι. που έχετε στα χέρια σας αυτό το τόσο δύσκολο εγχείρημα. Δύο ερωτήματα θέλω να σας θέσω. Το πρώτο ερώτημα είναι το θέμα των ε, νέων μορφών απομόνωσης. Έχω δει στην ε, Νότια Οσετία το νέο αυτό τείχος του Βερολίνου κατά κάποιο τρόπο. Έχετε κάνει αρκετά για να μπορέσετε να σταματήσετε αυτή τη διαδικασία. Δεύτερον, η Ρωσία είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός παράγων στο Νότιο Κάυκασο και όχι βέβαια ένας σταθεροποιητικός παράγων από τη δική μας οπτική γωνία. Είχε ένα αρνητικό ρόλο στη Γεωργία, υποχρέωσε την ε, Αρμενία να μην υπογράψει τη Συμφωνία για τον Αγκόνο Καραμπάχ. Το ερώτημά μου είναι, εάν έχετε την πρόθεση να αντιμετωπίσετε τη Ρωσία και με ποιο τρόπο, ποιο είναι το μήνυμα το οποίο θέλετε να δώσετε στη Ρωσία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Μάμικινς, ο οποίος είναι και ο εισηγητής μας για τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε εκπρόσωπε, θέλω και εγώ να εκφράσω την ε, ευγνωμοσύνη μου σε εσά για αυτά τα οποία μας έχετε παρουσιάσει και φυσικά για το έργο σας το οποίο δεν είναι καθόλου εύκολο, είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο και πολύπλοκο εγχείρημα. Δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε <clears throat> τη σημασία του έργου σας σε αυτή την τόσο δύσκολη περιοχή. Προσωπικά λοιπόν θέλω να σας ευχαριστήσω για την υποστήριξη που μου έχετε δώσει σε μένα προσωπικά ως εισηγητού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όταν προετοίμαζα την έκθεση για τη Γεωργία. Όλα αυτά ήταν πάρα πολύ χρήσιμα λοιπόν για μένα. Δύο ερωτήματα έχω. Καταρχήν, για τα κατεχόμενα εδάφη, την Αυχασία και την Νότια Οσετία μέσα στην επικράτεια της Γεωργίας. Με ποιο τρόπο θα μπορούσαν να γυρίσουν αυτά τα εδάφη και οι κατοικοί τους στον συνταγματικό χώρο, στη συνταγματική επικράτεια της Γεωργίας. Φυσικά η εδαφική ακεραιότητα της Γεωργίας είναι κάτι το οποίο κανείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να διαφυσβητήσει. Ένα δεύτερο ζήτημα. Τι είδους δυνατότητες, τι σενάρια βλέπετε για μια ενδεχόμενη συμφωνία που θα μπορούσε να συνάψει η Ρωσία με αυτά τα αποσχιστέντα εδάφη, την Απχασία και, Απχαζία και την Νότια αιτία Και τι κινδύνους βλέπετε να ελοχεύουν μέσα σε αυτές τις συμφωνίες. Κύριος Τένοκ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Σάλμπερ και πάλι <clears throat> τα συγχαρητήριά μου εξ ονόματο τη ομάδα ΙΣΙΑΡ των και μεταρρυθμιστών. Η ομάδα μου αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην περιοχή αυτή όπου δραστηριοποιείστε. Ε, σας εύχομαι κάθε επιτυχία καταρχήν για τη δυνατότητά σας να πάτε στον Αγκόνο Καραμπάχ, αλλά το Αζερβαϊτζάν δεν επιτρέπει σε κανένα ε, ακόμα και εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πάει σε αυτή την περιοχή. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς βλέπετε την κατάσταση σε σχέση με την συμμετοχή της Αρμενίας στην Ευρωασιατική Ένωση και τι σημαίνει αυτό και για το τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να κρατήσουμε την επαφή μας σε φιλικό επίπεδο με την Αρμενία παρά τις πιέσεις που υφίσταται για να ενταχθεί στη ρωσική τροχιά και δεύτερον πώς θα μπορούσε το Ναγκόνο Καραμπάχ να ενταχθεί σε αυτήν την ε, Ευρωασιατική <clears throat> ε, Ένωση. Είδαμε ήδη ότι το Καζακστάν έχει ήδη εμπλακεί μέσα στα πλαίσια της Ισλαμικής διάσκεψης με το Αζερμπαϊτζάν και τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκεί <clears throat> υλοποιούνται ή όχι. Ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο να επισκεφτείτε την περιοχή αυτή και επίσης υπήρχε μια αποστολή της ε, ΕΠΑ η οποία θα μπορούσε να αναπτυχθεί εκεί αν η ομάδα του Μίνς καταφέρει να εξασφαλίσει μια κίνηση προς μια ειρηνική διευθέτηση. Για το θέμα της γεωργίας. Φαίνεται ότι και η περιοχή του Λούγκατς και του Ντόμπασκ θα πάρει τη μορφή της Νότιας Οσετίας ή των άλλων περιοχών του Καυκάσου. Αυτή είναι κάπως η, φαίνεται η θέληση της Ρωσίας. Αλλά τα εδάφια αυτά που κατέχονται από τους Ρώσους η Απχαζία και η Νότια Οσετία έχουν πολύ λίγες ξένες επενδύσεις, πολύ ασθενικές οικονομίες. Μπορούμε να περιμένουμε, να περιμένουμε κάτι διαφορετικό στο Λουγκάν, στο Ντονέτσκ και στην Κρυμαία. Μπορούμε με τις χαμηλές τιμές του πετρελαίου να περιμένουμε ότι θα υπάρξει λόγω των κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μια ε, ένεση κονδυλίων στην Κρυμαία και την ε, Ανατολική Ουκρανία ή θα καταλήξουν να πάρουν τη μορφή που είδαμε να έχει πάρει η Νότια Οσετιακή Απκαζία τις τελευταίες δεκαετίες στη Γεωργία. Ο κύριος Νάρτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον κύριο Σάλμπερ, για την εξαιρετική παρουσία στην οποία έκανε και για τις ε, παρατηρήσεις τις συγκεκριμένες τις οποίες έκανε. Όταν βλέπω την κατάσταση όμως ε, στην Οσετία και στην ε, Απχαζία, θυμίζω ότι το Ναγκόρνο Καραμπάχ είναι εθνοτικά περίπου καθαρή περιοχή αλλά παρόλα αυτά έχει υπάρξει ουσιαστικά μια εκαθάριση φυλετική ε, στον διάδρομο ανάμεσα στη δημοκρατία της Αρμενίας και στο ίδιο το Άνω Καραμπάχ. Μιλάμε τώρα για εθνοκαθάρσεις και στην Οσετία και στην Αρχαζία και στην περιβάλλουσα γεωγραφική ζώνη του Άνω Καραμπάχ, οι οποίες διεξάγονται και σταθεροποιούνται σε χρόνο και ε, δημιουργούν μία de facto κατάσταση αντίστοιχη με την Ισραηλινή παρέμβαση στα ε, Παλαιστινιακά εδάφη. Εμείς βλέπουμε ότι υπάρχει μία στασιμότητα μέσα στην ε, σαπίλα ουσιαστικά και η κατάσταση χειροτερεύει συνεχώς. Δεν έχουμε δυνατότητες επίλυσης της κρίσης και ταυτόχρονα βλέπουμε ότι παραβιάζονται όλες οι αρχές του δικαίου. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Κύριε Ζάλμπερ, σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Εκ μέρους του ΕΛΚ υποστηρίζουμε πολύ την ε, Συμφωνία Σύνδεσης ε, Ένωσης και Γεωργίας και είχαμε την ευκαιρία πριν από μερικές εβδομάδες να συζητήσουμε τις προόδους που σημείωσε η Γεωργία στις μεταρρυθμίσεις της, το κράτος δικαίου κλπ. με τον Υπουργό Δικαιοσύνης τους. Κατά την ανταλλαγή εκείνη απόψεων είδαμε επίσης με μεγάλο ενδιαφέρον την πρόοδο που γίνεται για τον τερματισμό της επιλεκτικής δικαιοσύνης που όταν καμιά φορά από την προηγούμενη κυβέρνηση. Θα ήθελα όμως να μου πείτε πώς βλέπετε εσείς τις εξελίξεις σε αυτό το θέμα εκ μέρους της γεωργιανής κυβέρνησης και των δικαστικών της αρχών. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κύριε Σάλμπερ, λέει κυρία Πύρη, για την παρουσίασή σας. Έχω ένα ερώτημα για κάτι που συζητιέται αυτή τη στιγμή στη Γεωργία την ίδια τις τελευταίες δύο εβδομάδες, γιατί ήμουν εκεί την περασμένη και με εξέπληξε ότι δεν το αναφέρατε. Είναι η συνθήκη που προτείνει η Ρωσία με την Αμπχαζία. Για μένα Πρόκειται για μια σιωπηλή προσάρτηση της Αρχοαζίας. Προβλέπεται η δημιουργία κοινών στρατευμάτων, κοινέ δομές ε, εφαρμογής ε, ορισμένων ε, νομοθετημάτων και κοινό σύστημα υγείας. Θέλω λοιπόν να μου πείτε ποια είναι η θέση της Ένωσης για όλα αυτά και οι επαφές σας με τους με τις αρχές της Αμπχαζίας τι σας λένε ως προς αυτό το θέμα. Φανταζόμαστε τι θα σήμαινε και για την Νότια Οζετία μια ανάλογη συνθήκη. Για πέστε μας κι εσείς. Thank you, Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Ζάρμπερ, τα συγχαρητήριά μου για, την, για το διορισμό σας. Πρώτα απ' όλα, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με μια ιστορική αναδρομή. Όλοι μας θυμόμαστε την έκθεση Χάλια Ταλιαβίνη για τη Γεωργία. Την εποχή του πολέμου του 2008 και τις κατηγορίες οι οποίες διατυπώθηκαν για αυτούς οι οποίοι ξεκίνησαν αυτήν την αντιπαράθεση μετά από τα γεγονότα της Κρυμαίας, η εικόνα είναι πάρα πολύ σαφής πια. Και πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι η Ρωσία με την επιθετική της πολιτική που δίνει λαβή σε εθνοτική κάθαρση, είναι υπεύθυνη για όλα αυτά. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι ακόμα στο έδαφος της ε, Γεωργίας έχουμε χιλιάδες άτομα που έχει χρειαστεί να φύγουν από τις αιστείες τους από την Νότια Οσετία και την Απχαζία, εσωτερικά εκτοπισμένα άτομα. Αναρωτιέμαι λοιπόν για το πόσο αποτελεσματική είναι η πολιτική μας εκεί. Είπατε ότι εμείς δεν αναγνωρίζουμε την ε, ανεξαρτησία αυτών των κατεχομένων εδαφών δεν θα ήθελα να πω ότι είναι de facto αποσχιστήσεις περιοχές, γιατί είναι de facto κατεχόμενες. Και εμείς δεν πρέπει φυσικά να αναγνωρίσουμε μια τέτοια αποσκύρτησή τους. Ποιοι είναι οι λόγοι λοιπόν για τους οποίους η Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να αναγνωρίζει την, νότια, την ε, απόσχηση της Νοτίας ως και της Απχαζίας εμπλέκεται σε σχέδια και προγράμματα εκεί. Θα βοηθήσουμε εμείς τη Ρωσία να εξασφαλίσει την ειρήνη εκεί και θα ασκήσουμε, <clears throat> θα δώσουμε τη δυνατότητα στη Ρωσία να φέρει αυτά τα εδάφη πολιτικά, οικονομικά και στρατιωτικά πιο κοντά στην ε, Ρωσία. Κάτι αντίστοιχο βλέπουμε να είναι κίνδυνος να συμβεί στην Ανατολική, Νοτιοανατολική Ουκρανία και στην Κρυμαία. Και να έρθω τώρα στον Αγκόνο Καραμπάχ, στο Άνω ε, Καραμπάχ, την Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν, την μακρά διαμάχη που υπάρχει σε αυτή την περιοχή. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσουμε αυτή την διαμάχη, αλλά πρέπει να θυμόμαστε ότι η εθνοτική κάθαση αποτέλεσε ένα τμήμα αυτής της διαμάχης. Τι θα κάνετε λοιπόν ε, και τι θα δείτε ακριβώς, τι θέλετε να δείτε όταν μεταβείτε εκεί. Γιατί πρέπει να λάβετε υπόψη και τις δύο πλευρές της διαμάχης και να δείτε σε τι οφείλονται αυτές οι διαμάχες. Πιστεύω ότι έχετε μια πάρα πολύ πολύπλοκη εντολή. Εμείς βρισκόμαστε πολύ κοντά στην κύρωση της Συμφωνίας Σύνδεσης με τη Γεωργία και εγώ προσωπικά υποστηρίζω ιδιαίτερα την κύρωση αυτής της συμφωνίας. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω ότι εσείς ιδιαίτερα και όλες μας οι χώρες θα πρέπει να ασκήσουν πίεση στην κυβέρνηση της Γεωργίας για να αποφευθούν όχι μόνο τα δύο μέτρα και τα δύο σταθμά στις δικαστικές διαδικασίες, αλλά να αποφευθούν και οι προφανείς δυσκολίες οι οποίες μπορούν να προκύψουν σε βάρος της αντιπολίτευσης εκεί. Έχουμε την δικαστική δίωξη εναντίον του, προ, του προηγούμενου Προέδρου της Γεωργίας και τώρα μια τέτοια αντίστοιχη διαδικασία έχει κινηθεί εναντίον του κόμματός του, εναντίον ενός μεγάλου κόμματος αντιπολίτευσης. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το αποδεχτούμε σε μια χώρα με την οποία μας συνδέει μια εταιρική σχέση. Γι' αυτό θα πρέπει να κάνουμε ότι μπορούμε περισσότερο να ασκήσουμε πίεση στην κυβέρνηση της Γεωργίας για να σταματήσει τέτοιου είδους ενέργειες. Χωρίς μικρόφωνο και πάλι ο πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ λέει και κάτι άλλο το οποίο δεν ακούει κανείς βέβαια. Μία σύντομη ερώτηση. Μπορείτε να μας πείτε περισσότερα για την Ατζαρία. Η Ατζαρία είναι τμήμα της Γεωργίας και ποιος είναι ο ρόλος της οικογένειας Απασιτζέ στην περίπτωση αυτή της Αζαρίας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο κύριος Κάρβαρ, ο Ντέιβιτ Κάμερον ζήτησε να επεκταθεί προς τα Ουράλια η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, προς τις χώρες όπως η Γεωργία και η Αρμενία. Βλέπετε να υπάρχει μέλλον προς τα εκεί. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να σας συγχαρώ για το διορισμό σας. Η κατάσταση στη Γεωργία είναι ιδιαίτερος περίπλοκη. Εμείς είμαστε υπέρ της Συμφωνίας Σύνδεσης βέβαια, αλλά πριν ψηφίσουν για τη Συμφωνία Σύνδεσης, πριν φτάσουμε στην Ολομέλεια, θα ήθελα να μπορούσαμε να ξεκαθαρίσουμε προς τις γεωργιανές αρχές ότι θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικές και να μην χρησιμοποιούν με επιλεκτικό τρόπο το σύστημα της δικαιοσύνης, το δικαστικό σώμα. Να μην δείχνουν ότι υπάρχει ισχυρή επιθυμία για πολιτική εκδίκηση μέσα από τις δικαστικές και ανακριτικές διαδικασίες της βάρος της προηγούμενης κυβέρνησης. Αφού επικυρώσουμε τη Συμφωνία Σύνδεσης, ε, δεν θα είναι τόσο δεκτική απέναντί μας η γεωργιανή κυβέρνηση. Πρέπει λοιπόν να το διευκρινίσουμε αυτό και περιμένουμε και από εσά να βοηθήσετε κύριε Πρέσβη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η κυρία Γκόμες. Ευχαριστώ και τον κύριο Ζάλμπερ. Πολλοί πιστεύουν ότι η Απχαζία και η Νότια Οσετία ήταν ε, ένα πρόκριμα για αυτά τα οποία συνέβησαν στην Κρυμαία και για αυτά τα οποία θα συμβούν στον Ταμπάς. Τι πληροφορίες έχετε τώρα για την κατάσταση των πληθυσμών της Οσετίας και της Απραζίας; Την τελευταία φορά που είχα πάει εγώ στη Γεωργία επισκέφθηκα τα σύνορα με την Νότια Οσετία και μας έδωσαν πληροφορίες ότι δεν υπήρχαν και πάρα πολλοί πληθυσμοί εκεί γιατί πολλοί είχαν φύγει και η κατάσταση χειροτέρευε στη Νότια Οσετία επιμένω ε, πάρα πολύ. Ε, τι πληροφορίες έχετε εσείς. Αυτή η απόσχηση στην ουσία οδήγησε στην απομάκρυνση του πληθυσμού ή έχει αρχίσει και επιστρέφει. Τι ακριβώς συμβαίνει. Τώρα για την συμφωνία που διαπραγματευόμεθα με τη Γεωργία την υποστηρίζουμε φυσικά και κατανοούμε τη σημασία της. Αλλά το θέμα της ανεξαρτησίας του δικαστικού σώματος είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό, καθοριστικό θα έλεγα. Και εγώ όταν είχα πάει εκεί είχα ανησυχήσει για τα στοιχεία τα οποία είχαμε συναντήσει. Δεν ξέρω τι κάνει η παρούσα κυβέρνηση. Τώρα για το Άνω Καραμπά απευθύνω έκκληση να συνεχίσετε να επιμένετε για επισκέψεις στο Άνω Καραμπάχ. Και ίσως θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε και κάποιον ανώτερό σας, τον είπα το εκπρόσωπο σαν παράδειγμα, έτσι ώστε να μεταφέρει τις διαμαρτυρίες σας προς την κυβέρνηση της, του Αζερμπαϊτζάν για τις δυσκολίες αυτές που δημιουργεί. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στις ερωτήσεις με τη σειρά με την οποία τέθησαν. Η πρώτη αφορούσε τα διαχείριση των συνόρων μεταξύ Αμπχαζίας και Νότιας Οσετίας και τη δράση της κυβέρνησης της Τυφλίδας. Αν έχουμε κάνει αρκετά για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Νομίζω ότι αυτό υπήρχε και πριν αναλάβω εγώ ο κάθε καινούργιος εκπρόσωπος που πήγαινε εκεί απέφτεινε κλήσεις σε όλες τις πλευρές και επιτόπου και από εδώ από τις Βρυξέλλες έγιναν προσπάθειες να πιστούν οι πλευρές να διευθετήσουν αυτό το θέμα του διοικητικού συνόρου και στον ΟΑΣΕ έχουν γίνει ανάλογες δηλώσεις. Έγιναν λοιπόν πολιτικές προσπάθειες τουλάχιστον να περιοριστεί αυτό το πρόβλημα. Ξέρουμε όμως ότι συνέχισε η συνοριοποίηση αυτή, το ξέρουμε. Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν και σειρματοπλέγματα και είναι πιο δύσκολη η πρόσβαση γενικά. Δεν μπορεί λοιπόν κανείς να πει ότι οι προσπάθειες να λυθεί το πρόβλημα ήταν επιτυχής, αλλά τουλάχιστον δεν έχουν χειροτερέψει. Δεν έχουν όμως φραγίσει όλα τα σύνορα. Η διαδικασία αυτή λίγο πολύ τελείωσε. Είναι δύσκολο να πει κανείς αν ο δρόμος της Ένωσης, που ακολούθησε η Ένωση ήταν αρκετά επιτυχής αλλά τουλάχιστον έγινε μια σοβαρή προσπάθεια να επηρεαστούν να αλλάξουν τα πράγματα και ακούστηκε η φωνή μας στη Μόσχα. Το δεύτερο θέμα ήταν, σχετιζόταν με τη Ρωσία ως σημαντικό παράγοντα στον Κάυκασο. Τι μήνυμα δίνουμε στη Ρωσία. Το μήνυμά μας στη Ρωσία Μήνυσα με τον Υφυπουργό Εξωτερικών Καράσιν είτε είναι να μας βοηθήσει να προχωρήσουμε επικοδομητικά στις συζητήσεις των, της Γενέβης. Το θεωρούμε δηλαδή πολύτιμο σύμμαχο. Σε μερικές περιπτώσεις αυτή η προσέγγιση λειτουργεί, σε άλλες όχι, όχι σε όλες. Υπάρχουν τα συμφέροντα, υπάρχουν μερικά συμφέροντα που τα παρακολουθούμε και εμείς και εκείνοι στενά αλλά το κύριο μέσα με μήνυμα είναι ας είμαστε όλοι επικοδομητικοί στον Κάφκασο. Τις τελευταίες εβδομάδες από τότε που παρακολουθώ τα πράγματα ακόμη στενότερα η Ρωσία έχει παίξει εκπληκτικά περιέργως επικοδομητικό ρόλο ιδίως ως προς τις συζητήσεις της Γενέβης και μεγαλύτερη συνεργασία υπήρξε με τη Ρωσία αλλά θυμίζω και τις συζητήσεις που γίνονταν επί μήνες μεταξύ του Υφυπουργού Καράσιν από τη μία και του ειδικού εκπροσώπου του Προέδρου της Γεωργίας για τις διμερείς σχέσεις τον κύριο Αμπάσιτζε από την άλλη. Κατάφεραν να κάνουν μερικά πράγματα στο σε εμπορικά θέματα, μεταφορές, που καρποφόρησαν. Και οι σχέσεις Γεωργίας-Ρωσίας προχώρησαν περιέργως καλά σε σύγκριση τουλάχιστον με αυτά που γίνονται στην Ουκρανία. Έχω λοιπόν την εντύπωση ότι το σχέδιο αυτό συμφωνίας της Ρωσίας με την Αμπχαζία είναι διαφορετικό θέμα και θα το συζητήσω γι' αυτό αργότερα. Τώρα για το ερώτημα του κυρίου Μαμίκιν πώς να επανέλθουν οι αποσχιστικές, οι αποσχισμένες περιφέρειες στη Γεωργία. Αυτό είναι πολύ δύσκολο θέμα και μακροπρόθεσμο. Το μόνο που θα μπορούσε να γίνει αν δεν υπάρξουν αναπάντεχες ιστορικές εξελίξεις θα ήταν η Γεωργία να καταργήσει ο Άρη ορισμένους φραγμούς που έθεσε μετά τον πόλεμο και που θα ήταν σοφότερο τώρα να αρχίσει να τα, τους καταργεί για να μπορούμε να πούμε ότι άλλαξαν οι νοοτροπίες. Στην Αμπχαζία πολλοί θέλουν να κρατήσουν ζωντανή την επικοινωνία με τη Γεωργία. Ενώ δυστυχώς αυτό που γίνεται μάλλον είναι κυρίως απομόνωση και απόρριψη. Μερικές φορές βέβαια δεν βοηθάει η πολιτική της Γεωργίας, ιδίως αυτά που είπε τελευταία ο Πρωθυπουργό ας πούμε. Αν μπορούσαν να μιλήσουν και αυτοί πιο ήπια, καλό θα ήταν. Το επόμενο ερώτημα αφορούσε το ρόλο της Αρμενίας και τι θα μπορούσε να γίνει για να πλησιάσει προς την Ευρώπη. Στην Αρμενία πολλοί θέλουν να κρατήσουν δεσμούς με την Ευρώπη. Μέχρι τώρα στις συνομιλίες που είχαμε τον πρόεδρο και τον πρωθυπουργό αλλά και άλλους από την κυβέρνηση βλέπω καθαρά ότι δεν είναι επιλογή αυτή αλλά ο μόνος τρόπος για την ανάπτυξή τους θα θέλουν να κρατήσουν δεσμούς με την Ευρώπη και είναι και διατεθειμένοι να κάνουν και κάτι πρακτικά γι' αυτό. Προς το παρόν βέβαια η Ρωσία έχει τη μεγαλύτερη επιρροή και δεν έχουν άλλη επιλογή οι Αρμένοι από το να μπουν στην Ευρωασιατική Ένωση. Όσο για το ορεινό Καραμπάχ και εκεί ζητάμε να παραμείνουν οι επαφές θα ήταν όμως αδύνατο να επιβάλλουμε οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή λόγω των εξελίξεων. Εμείς θέλουμε οι συνεννοήσεις να γίνονται αλλού, ας πούμε εδώ στις Βρυξέλλες. CSDP, η ειρηνευτική επιχείρηση του ΑΣΕ. Θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά θα χρειαζόταν μεγάλη εφευρετικότητα και η οποία δεν προβλέπεται αυτή τη στιγμή. Πρέπει να το σκεφτούμε όμως την κατάλληλη στιγμή όμως. Στην Αμπχαζία και την Νότια Οσετία η οικονομία εκεί είναι πολύ, σε πολύ άσκημη κατάσταση. Από πολλές επισκέψεις μου εκεί δεν μπορώ να πω ότι είναι χειρότερη από άλλες κοντινές γειτονικές περιοχές στην Αρμενία ή στην Ήπεθρο της Γεωργίας. Υπάρχουν πολλές επενδύσεις ρωσικές εκεί, ιδιαίτερα στην Νότια Οσετία. Φαίνεται ότι γίνονται πολλά στις υποδομές στην πόλη ή μάλλον το χωριό του Σκινβάλι, δεν είναι πραγματικά πόλη, πολλές οικοδομές και δεν θα έλεγα, ότι, η κατάσταση, δεν ότι η κατάσταση εκεί είναι πολύ χειρότερη από ό,τι σε ορισμένα σε άλλε περιφέρειες, ιδίω στην Ήπεθρο. Σε πολλά ερωτήματα υπήρχε το θέμα της λεγόμενης επιλεκτικής δικαιοσύνης στη Γεωργία. Αυτό δεν αφορά άμεσα τη δική μου εντολή αλλά τα εσωτερικά της γεωργίας και γι' αυτό όταν συζητάμε αυτό το θέμα με τους γεωργιανούς αφήνω την πρωτοβουλία στην αντιπροσωπεία μας στην Τυφλίδα. Πάντως όταν έχω επαφές δεν αφήνω καμία αμφιβολία ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σοβαρές αμφιβολίες για τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται πολλές φορές η δικαιοσύνη, ιδίω προς τους προηγούμενους ηθήνοντες. Τώρα για την συνθήκη της Ρωσίας με την Αμπχαζία. Δίκιο έχετε, έπρεπε να το είχα πει από την αρχή. Ας τα πω όμως τουλάχιστον τώρα. Πρόκειται όντως για σιωπηλή προσάρτηση Ξέρουμε ότι η Γεωργία λέει, χρησιμοποιεί τέτοια ορολογία. Αλλά αν δούμε αυτή τη συνθήκη, μιλάει για, ένα για εναρμόνιση νομοθεσίας και άλλους κανόνες, για ολοκλήρωση μιλάει, αλλά δεν νομίζω ότι μπορούμε να μιλήσουμε για προσάρτηση. Αν εφαρμοστεί όπως γράφεται ότι θα εφαρμοστεί. Υπάρχει όμως και μια αμπχαζική αντιπρόταση που μειώνει, μειώνει, νερώνει πολλά από αυτά που είχε η αρχική ρωσική πρόταση. Τώρα δεν γίνεται λόγος για στρατηγική εταιρική σχέση. Αλλά έχουν αφαιρεθεί πολλά, πολλές ρήτρε για στρατιωτική συνεργασία και γι' αυτό η πρώτη μας ανάλυση αυτής της αντιπρότασης είναι ότι μειώνει το βαθμό σύγκλησης Ρωσίας-Αμπχαζίας πλησιάσματος. Δεν ξέρουμε τι τελικά θα γίνει, με τι μορφή θα υπογραφεί αυτή η συνθήκη, γιατί φανταζόμαστε ότι θα υπογραφεί φέτος, μα πριν τελειώσει ο χρόνος. Διότι έχει πολύ σχέση με χρηματοδότηση από τη Ρωσία για την περιοχή αυτή. Α δούμε όμως. Προς το παρόν Είπαμε στους Γεωργιανούς ότι θα δούμε και εμείς και εκείνοι ποια θα είναι η τελική εκδοχή της συνθήκης. Θα συζητηθεί ακόμη το πράγμα και στην Αμπχασία αλλά και από τις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία και την Αμπχαζία και τότε θα δούμε τι σχόλια θα κάνουμε. Φυσικά λέμε και στους Απχάζιους και στους Ρώσους ότι η υπογραφή της συμφωνίας όπως την προτείνουν οι Ρώσοι μας θέτει πολλά προβλήματα διότι ως προς το τι θα παραμείνει από την Απχαζική κυριαρχία μετά την εφαρμογή αυτής της συμφωνίας. Το είπα αυτό και στον Υφυπουργό Καράσιν αλλά και στον de facto Υπουργό Εξωτερικών Υπουργό Εξωτερικών της Αμχαζίας τον κύριο Τσιρίκμπαν. Πολλές φορές το θίξαμε αυτό το θέμα. Αυτό νομίζω απαντάει και για το θέμα με τις επαφές με την Απχαζία. Σε συνεχή διάλογο βρισκόμαστε, όχι καθημερινό, αλλά συνεχή. Έχουμε μετά το θέμα του κατά πόσον, έτσι διατυπώθηκε τουλάχιστον πιστεύω, αν θα πρέπει να βοηθήσουμε τους Απχαζίους, αλλά αν κάνοντας αυτό ε, έμεσα βοηθούμε τους ε, Ρώσους να εδραιώσουν την κατοχή της Απχαζίας. Νομίζω ότι αυτό το οποίο κάνουμε, το να έχουμε σχέδια ανάπτυξη στην περιοχή και να κρατήσουμε ζωντανή την επαφή με την περιοχή αυτή, σίγουρα δεν βοηθούμε τους ηγέτες της Απχαζίας και δεν βοηθούμε τη Ρωσία αυτού, αυτοί που προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε είναι η κοινωνία των πολιτών της Απχαζίας. Και μπορώ να σας πω ότι έχουμε πολλές επαφείς που μας δείχνουν ότι υπάρχουν πολλοί στην Απχαζία που δεν θεωρούν ότι ο τελικός στόχος τους θα πρέπει να, είναι, να γίνει η Απχαζία τμήμα της Ρωσίας. Πολλοί από αυτούς λοιπόν θα θέλαν να διατηρήσουν τη δική τους ε, κυριαρχικότητα και ανεξαρτησία. Ο κύριος Τσερίκ Μπάρο facto Υπουργός Εξωτερικών, είναι ένα από τα, κατά κάποιο τρόπο, από αυτούς οι οποίοι ε, κίνησαν τη διαδικασία για να υπάρξουν κάποιες τροποποιήσεις στη Συμφωνία Απχασίας-Ρωσίας. Δεν θέλουμε λοιπόν να βοηθήσουμε την ηγεσία της Απχασίας ούτε τη Ρωσία. Θέλουμε να βοηθήσουμε όμως την κοινωνία των πολιτών εκεί με τον απότερο στόχο να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την ε, επανενσωμάτωση αυτών των εδαφών στην ε, Ρωσία, διότι εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζουμε την εδαφική ακεραιότητα της Γεωργίας. Ένα άλλο ερώτημα που τέθηκε <clears throat> είναι το αν η Γεωργία μπορεί εν καιρό να είναι υποψήφια για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορώ να σας δώσω καμία <clears throat> απάντηση. Ξέρουμε ότι οι Γεωργιανοί θέλουν να πλησιάσουν την Ευρώπη, εργάζονται για να μπορέσουν να το κάνουν αυτό πραγματικότητα. Το κατά πόσον όμως σε τελική ανάλυση θα θέλουν να είναι υποψήφιοι για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό δεν είναι σαφές προς το παρόν. Αυτή τη στιγμή δεν είναι υποψήφια η χώρα αυτή. Ετέθη το θέμα της Ατζαρίας. Εγώ πήγα μια φορά εκεί ως ε, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρουμε ότι μετά από την ε, ε, μεταπολίτευση στην Γεωργία, η Ατζαρία επανήλθε μέσα στην Γεωργία. Η Γεωργία έχει υποσχεθεί να διατηρήσει αυτή την αυτονομία της Ατζαρίας. Αυτά όμως τα οποία βλέπουμε μέχρι στιγμής είναι ότι δεν υπήρξε πραγματικά μία τήρηση αυτής της υπόσχεσης. Αν δούμε λοιπόν την ε, επίπτωση που μπορεί να έχουν αυτά τα γεγονότα της Αζαρίας στην Οσετία και την, ε, στην Νότια Οσετία και την Απχαζία, αν θέλουν να επανέλθουν στην Γεωργία, φυσικά δεν αποτελεί το καλύτερο παράδειγμα για τις περιοχές αυτές. Το ερώτημα είναι αν η Απχασία και η Νότια Οσετία ήταν ουσιαστικά το παράδειγμα για αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα στον Τόνες και στην, στο Λουγκάνσκ στην Ουκρανία. Δεν είμαι σίγουρος ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει. Βέβαια θα μπορούσε κανείς πάντα να το ερμηνεύσει με αυτόν τον τρόπο. Όταν συναντήθηκα με την ηγεσία των Αζέρων του Αζερβαϊτζάν μας μου είπανε ότι αν είναι κάποιος μέρος της, ε, των, χωρών που θέλουν να πλησιάσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση κινδυνεύει κανείς να χάσει την εδαφική του ακαιρεότητα. Εγώ δεν πιστεύω ότι πρέπει να το δούμε έτσι το θέμα αυτό. Πιστεύω σε μεγάλο βαθμό είναι ακόμα ανοιχτέ οι και οι εξέλιξεις. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε κατά πόσον όλες αυτές οι συνθήκες είναι συγκρίσιμες προς το παρόν δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτά τα οποία γίνονται στην Ουκρανία είναι χαλκομανία αυτών που έχουν γίνει στη Γεωργία. Πιστεύω ότι όλες αυτές οι συγκρούσεις και οι διαμάχες έχουν τις ιδιαιτερότητές τους και πρέπει να λάβουμε υπόψη πάρα πολύ προσεκτικά τις ιδιαιτερότητές τους. Κάτι το οποίο είναι σαφές όμως είναι ότι η Ρωσία προσπαθεί να εξασφαλίσει ότι θα διατηρήσει την επιρροή της σε αυτή την περιοχή που φυσικά είναι πολύ σημαντικό στοιχείο της ε, πρώην Σοβιετικής Ένωσης και ξέρουμε πώς θα αντιμετωπίζει αυτά ο πρόεδρος Πούτιν. Για τα άτομα τα οποία βρίσκονται και στις ε, de facto οντότητες οι οποίοι αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι αυτών των οντοτήτων περισσότερα προβλήματα από στο παρελθόν. Εγώ ξέρω κάπως την κατάσταση στη Νότια Οσετία. Είχα επισκεφθεί την περιοχή αυτή πριν από το 2008. Δεν νομίζω ότι είναι χειρότερα τα πράγματα από ό,τι παλαιότερα. Ίσως και λόγω ακριβώς της έντονης παρουσίας χρημάτων από τη Μόσχα τα πράγματα να είναι καλύτερα. Αλλά το να πούμε ότι ζουν χειρότερα από ό,τι στο παρελθόν αυτό δεν θα ήταν δίκιο. Μια τελευταία παρατήρηση αναφέρεται πάντα στο Άνω Καραμπάχ. Γιατί το έτοιμά σα να συνεχίσω να ετούμε την παρουσία μου στην περιοχή αυτή. Φυσικά και θα το κάνω αυτό και πάντα έχω την ελπίδα ότι σε ένα έλογο χρονικό διάστημα θα γίνει η ελπίδα αυτή πραγματικότητα και θα επισκεφθώ το Άνω Καραμπάχ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίασή σας. Ερχόμαστε στο επόμενο σημείο της σημερινής διάταξης, που είναι το θέμα της Συμφωνίας Σύνδεσης. Ο κύριος Μάμικινς είναι ο εισηγητής μας εδώ και θα πρότεινα τα σημεία 5 και 6 θα τα συζητήσουμε από κοινού. Μπορώ να ζητήσω από κάποιον συνάδελφο να αναλάβει την Προεδρία. Κόουσο. Eh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ξεκινώντας θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους κοιόδης εισηγητές για τη σύνδρομή τους και όλους τους ευρωβουλευτές συναδέλφους οι οποίοι υπέβαλαν τις δικές τους τροπολογίες. Τις διάβασα προσεκτικά νομίζω και θεωρώ ότι είναι σημαντικές συνεισφορές με στόχο την βελτίωση της συγκεκριμένης πρότασης. Τα σχόλιά σας λοιπόν συνάδελφοι είναι σημαντικά και σας διαβεβαιώ ότι θα βοηθήσουν έτσι ώστε να καταλήξουμε σε μια καλή συμβιβαστική και εξισορροπημένη έκθεση. Η εντύπωσή μου είναι ότι η έκθεση αυτή θα μπορέσει να βοηθήσει την Γεωργία να έλθει πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε επίπεδο οικονομικό και σε επίπεδο πολιτικό. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής θα έλεγα και ικανοποιημένος γιατί και η δική μου βασική θέση την οποία ε, προτείνω στην έκθεση είναι να στηρίξουμε την άποψη που λέγει ότι πρέπει η Γεωργία να έρθει ακόμα πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι προσπαθούμε ε, να εκφραστούμε θετικά για τις μεταρρυθμίσεις οι οποίες έχουν συμβεί στην Γεωργία στα πλαίσια της προπαρασκευής για την ε, συμφωνία αυτή ε, τη Συμφωνία Συνεργασίας. Θα ήθελα επίσης όμως να μην παραλείψουμε να υπογραμμίσουμε το εξής. Αυτό το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε με την έννοια της επιλεκτικής απόδοσης δικαιοσύνης υπάρχει και στην έκθεσή μου και στις δικές σας τροπολογίες. Έχω την εντύπωση ότι δεν μπορούμε εμείς να δουλέψουμε ε, στη θέση της Γεωργίας για να αλλάξουν τα πράγματα. Τη δουλειά αυτή πρέπει να την κάνουν οι ίδιοι οι Γεωργιανοί το ίδιο το δικαστικό σώμα της χώρας θα πρέπει να ξεκινήσει κάποιες αλλαγές και κάποιες μεταρρυθμίσεις. Εάν βέβαια πολιτικοποιηθούν οι αλλαγές αυτές οι αναμενόμενες, τότε αυτό θα δυσκολέψει την κατάσταση ακόμα περισσότερο. Ε, νομίζω ότι και στη δική μου χώρα το δικαστικό σώμα πέρασε και αναφέρομαι στη Λετωνία πέρασε από τις διαδικασίες αυτές της μεταρρύθμισης μετά από κάποιες σημαντικές αλλαγές στη χώρα. Ε, και νομίζω ότι έχουν προχωρήσει τα πράγματα στην Γεωργία ίσως και περισσότερο από αυτά τα οποία έχουν συμβεί στη δική μου χώρα, λέει ο κύριος Μαμίνκινς. Το κράτος δικαίου λοιπόν είναι ένα θέμα στο οποίο ε, γίνονται ορισμένα σχόλια και από πλευρά σας και είναι σαφές ότι θα πρέπει εδώ οι απόψεις νομικών νομομαθών και εμπειρογνωμόνων να μας διαφωτίσουν ακόμα περισσότερο. Πάντως επανέρχομαι σε αυτό που είπα πριν. Το ανεξάρτητο δικαστικό σώμα είναι, είναι πραγματικά το σημείο πάνω στο οποίο θα θεμελιωθεί η δημοκρατία στη χώρα. Τώρα για το ρόλο της Ρωσίας και την επιρροή της Ρωσίας στις συγκεκριμένες αυτές διαδικασίες. Σαν εισηγητής θα ήθελα να πω ότι πράγματι θα πρέπει να δώσουμε προσοχή στην γεωργία και να βοηθήσουμε την γεωργία παρά να ασχολούμαστε και να κατηγορούμε και να υπογραμμίζουμε τον αρνητικό ή όχι ρόλο της Ρωσίας και την παρέμβασή της στην γεωργία είναι δύσκολο για την Γεωργία να σταθεί στα πόδια της μετά από τον πόλεμο του 2008. Όταν έκανα την αρχική μου πρόταση πάντα έμεινα στα της Γεωργίας και δεν ήθελα να αφιερώσω το χρόνο και την ενέργειά μου στην Ρωσία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μάνικενς. Κύριο Στετίνα, έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να χρησιμοποιήσω τη μετική μου γλώσσα για να γίνω σαφέστερος. Το ΕΛΚ υποστηρίζει την κύρωση της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Γεωργίας Πιστεύουμε θα είναι θετικό αυτό για την ε, γεωργία και τους πολίτες της, θα πλησιάσει τη χώρα αυτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα ενισχύσει τις κοινέ αρχές και αξίες. Με τον τρόπο αυτό θέλουμε ένα σαφές μήνυμα από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, λαμβάνοντας υπόψη τον ε, ακήρυκτο πόλεμο που ισχύει αυτή τη στιγμή στα ανατολικά και νοτιοανατολικά σύνορα της Ουκρανίας από τους Ρώσους και στην Απχαζία και Νότια Οσετία που έχουν αποσχίσει. Βλέπουμε τώρα ότι υπάρχουν και συμφωνίες για μια περαιτέρω ολοκλήρωση και ενσωμάτωση, όπως έχει αναφερθεί. Θα πρέπει λοιπόν των περιοχών αυτών στην Ρωσία. Θα πρέπει να κάνουμε λοιπόν ό,τι μπορούμε για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την ε, διαδικασία αυτή προσέγγισης και τη συμφωνία σύνδεσης. Θέλω συγχαρώ τον κύριο Μάνικινς για την ε, έκθεσή του, για το γεγονός ότι πήγε προσωπικά στην Γεωργία και μίλησε με όλους τους υπεύθυνους εκεί και ο ίδιος και εγώ ήδη πρωτού πάμε στην, μπούμε στον πολιτικό στίβο ήμασταν δημοσιογράφοι στην Γεωργία και έχουμε λοιπόν κοινό έδαφος ως εκ τούτου και χαίρομαι που οι τροπολογίες θα μας επιτρέψουν να αντιμετωπίσουμε τα πιο κέρια και καυτά θέματα, συγκεκριμένα τα θέματα της κατάχρησης της δικαστικής εξουσίας για να υπάρξει αντεκδίκηση στο πολιτικό επίπεδο. Αυτό έχει αναφερθεί πολλές φορές λοιπόν στη συζήτηση αυτή από εκπροσώπους πολλών πολιτικών δυνάμεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Κάτι ακόμα το οποίο για μένα ήταν ιδιαίτερα οδυνηρό. Το 1968 μπήκαν οι Σοβιετικές δυνάμεις και κατέλαβαν την Τσεχοσλοβακία. Γιατί σας το λέω τώρα αυτό. Γιατί η κομμουνιστική ηγεσία στη χώρα μου χρησιμοποίησε την εφημιστική διατύπωση είσοδος των στρατευμάτων του Συμφώνου της Βαρσοβίας. Εμείς ξέραμε όμως ότι αυτό ήταν μια καθαρή κατοχή. Δεν θελήσαμε να χρησιμοποιήσουμε μια τέτοια διατύπωση. Και σας τα λέω αυτά γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι μπορούν να θέλουν να χρησιμοποιήσουν κάπως ε, καλοπιστικές εκφράσεις, να μην μιλάνε για κατοχή των εδαφών, αλλά για περιοχές που είναι υπό απόσχηση κτλ. Γι' αυτό εγώ θέλω να τονίσω ότι θα πρέπει να παραμείνουμε στη διατύπωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2011 όταν ελέγχθη ότι πρόκειται για καθαρή κατοχή των εδαφών αυτών. Υπάρχει και το θέμα της φιλελευθερωποίησης για τις προξενικές θεωρήσεις. Η Κομισιόν μας είπε την προηγούμενη εβδομάδα ότι η Γεωργία εκπληρεί τις προϋποθέσεις για την πρώτη φάση φιλελευθερωποίησης προξενικών θεωρήσεων, περνάνε τώρα στη δεύτερη φάση, η οποία εν καιρό θα μας φέρει στην δυνατότητα να έχουμε ε, ελεύθερη διακίνηση χωρίς βίζα. Και απλώς το αναφέρω αυτό λόγω επευκαιρία. Κύριε Μάμκινς, λοιπόν, προσβλέπω στο να καταθέσω ε, τροπολογίες συμβιβασμού και να συναντηθώ μαζί σας την επόμενη εβδομάδα. Ελπίζω θα μπορέσουμε να βρούμε λοιπόν τον χρόνο για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια τελική διατύπωση και εξ ονόματος του ΕΛΚ θέλω και πάλι να τονίσω την θέλησή μας, την αποφασιστικότητά μας για να γίνουν όλες οι απαραίτητες προσπάθειες για την καλή προετοιμασία αυτής της έκθεσης. La palabra, señor um, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ θα είμαι πολύ σύντομος. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τον προλαλήσαντα και τον κύριο Μάμικινς. Ε, νομίζω ότι είναι πολύ καλό το κείμενο όσο έχει παρά τις πολλές τροπολογίες. Οι περισσότερες αφορούσαν το θέμα της επιλεκτικής δικαιοσύνης. Η πράσινη συνήθως είναι υπέρ μιας σαφούς διατύπωσης, αλλά σε αυτή την περίπτωση θα ήθελα να σας συστήσω φρόνηση για τις τροπολογίες τους, διότι το να λέμε ότι η επιλεκτική δικαιοσύνη είναι το μόνιμο και μόνο πρόβλημα, ενώ ξέρουμε ότι υπήρξαν και επιτυχίες στις δικαστικές μεταρρυθμίσεις, δεν βοηθάει και πολύ τη γεωργία. Θα προσπαθήσουμε να τα συμβιβάσουμε αποφεύγοντας τη συνεχή χρησιμοποίηση του όρου επιλεκτική δικαιοσύνη. Κατά τα άλλα το κείμενο νομίζω είναι πολύ καλό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα δύο σημεία κυρίως ε, να υπογραμμίσω. Καταρχάς η έκθεση είναι καλή έκθεση. Γενικά το λέω αυτό. Και χρησιμοποιεί αν θέλετε και ε, τον κοινοβουλευτικό λόγο που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί από το κοινοβουλίο μας στο παρελθόν. Θα ήθελα να πω όμως εδώ ότι αυτό που έχει σημασία είναι να μιλήσουμε και για τη Ρωσία στην έκθεση αυτή. Η παρούσα κατάσταση φυσικά και συνδέεται με τις ενέργειες της Ρωσίας και με τις υποχρεώσεις που ανέλαβε η Ρωσία μετά από την ειρηνευτική συμφωνία ή μάλλον τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός του 2008 και θα πρέπει η Ρωσία χωρίς καμία εξαίρεση να σεβαστεί τις υποχρεώσεις και να παράσχει απεριόριστη πρόσβαση στην ομάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις περιοχές τις οποίες κατέχει. Και θα πρέπει επίσης να ανακαλέσει την αναγνώριση της Νότιας Οσετίας και της Απχαζίας. Αυτό ζητά ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου. Θα υποστηρίξω επίσης και την καταδίκη της λεγόμενης borderization, δηλαδή σε εισαγωγικά το βάζουμε συνοριοποίησης. Τώρα να έλθω στο θέμα της επιλεκτικής δικαιοσύνης στην Γεωργία. Εγώ θα υποστηρίξω την χρήση του συγκεκριμένης αυτής φράσης. Προέρχομαι από μια χώρα η οποία πέρασε από μια μακρά περίοδο μεταρρύθμισης του δικαστικού. Και γι' αυτό ακριβώς ε, οι εταίροι μας θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν την ευκαιρία την οποία έχουν για να ε, καταλήξουν σε μια κάποια θετική λύση. Σαν Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε ξεκαθαρίσει εμείς το πού είναι το πρόβλημα πριν ε, επικυρώσουμε την συμφωνία αυτή την οποία φυσικά και θα υποστηρίξω. Διευκρινίσαμε λοιπόν προς τις Γεωργιανές Αρχές πως οφείλουν να είναι πάρα πολύ προσεκτικές και να μην χρησιμοποιούν ε, την επιλεκτική δικαιοσύνη και να μην δίδουν την απαράδεκτη εντύπωση ότι εκδικούνται ε, τους πολιτικούς τους αντιπάλους. Αυτή η αίσθηση της ύπαρξης επιθυμίας για πολιτική εκδίκηση είναι κάτι το οποίο φύγει το αντικειμενικό των δικαστικών και ανακριτικών διαδικασιών. Ευχαριστώ κύριος Γιούρεκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η προετοιμασία αυτής της έκθεσης νομίζω ότι είναι πάρα πολύ θετική για, την, ε, για να αποτελέσει βάση για τη συζήτηση για τα θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης Γεωργίας. Και συμμερίζομαι την κύρια την κεντρική ιδέα αυτής της έκθεσης και πρέπει να το πω αυτό εξ ονόματος συντηρητικής ομάδος ότι εμείς υποστηρίζουμε το ταχύτερο δυνατό να συναυτεί αυτή η συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γεωργίας. Θέλουμε να δώσουμε όλη μας την υποστήριξη για να υπάρξει δημοκρατικοποίηση στη Γεωργία και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα γίνουν παρεμβάσεις οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν ως αποτέλεσμα όλες οι μεταρρυθμίσεις οι οποίες έχουν γίνει μετά από την ε, επανάσταση των Ρόδων να τεθούν εν αμφιβόλο. Γιατί η προηγούμενη κυβέρνηση έχει καταφέρει να προχωρήσει αυτές τις μεταρρυθμίσεις και, το, και η τωρινή κυβέρνηση. Θέλουμε λοιπόν η διαδοχή στην εξουσία να γίνεται με ένα ομαλό τρόπο, αλλά στην περιοχή αυτή είναι πολύ δύσκολο να γίνεται πραγματικότητα. Κοιτάξτε τι έγινε στην Ουκρανία, πόσο δύσκολο ήταν για την Ουκρανία να αλλάξει κυβέρνηση. Πιστεύω λοιπόν ότι με τον τρόπο αυτό μπορούμε να ελπίσουμε να πάνε τα πράγματα κάπως καλύτερα στην ε, ε, Γεωργία. Ε, σε τι τώρα εγώ θέλω να δώσω έμφαση Στι τροπολογίες μου. Πρέπει να λάβουμε υπόψη την ανάγκη συνένεσης όλου του πληθυσμού της Γεωργίας για να υπάρξει μια προσέγγιση προς την Ευρώπη και προς την ευρωατλαντική διάσταση. Δεν πρέπει λοιπόν να ξεχάσουμε αυτή την βασική οδηγό ιδέα, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική για την κοινωνία της Γεωργίας. Δεύτερον, Το σύνθημά μας και το οδηγό μας νήμα σε ό,τι αφορά τη σχέση μας με τη Γεωργία εναντί της Ρωσίας θα πρέπει να είναι η αλληλεγγύη. Θα πρέπει να βοηθήσουμε όλες αυτές τις χώρες οι οποίες προήλθαν από την αποσύνθεση της Σοβιετικής Αυτοκρατορίας. Μία ιστορική παρένθεση, αν μου επιτρέπετε. Περίπου πριν από 100 χρόνια, μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, φαινόταν ότι η ρωσική αυτοκρατορία θα προχωρούσε σε μια διαδικασία από απεικιοποίησης διότι περί αυτού πρόκειται. Ακολούθησε όμως μια σειρά από επαναστάσεις, η Ρωσική Επανάσταση και άλλες επαναστάσεις που ουσιαστικά πάγωσε αυτή τη διαδικασία. Μόνο τώρα μπορούν αυτές οι χώρες να αποκτήσουν την ελευθερία τους. Έχουν χαθεί 100 χρόνια στο δρόμο προς την ελευθερία. Ήταν ιδιαίτερα δυναμική η διεκδίκηση της ελευθερίας στις χώρες αυτές, αλλά στραγγαλίστηκε από την ρωσική αρκούδα. Πρέπει λοιπόν εμείς να υποστηρίξουμε όλες αυτές τις χώρες και να ζήσουμε μαζί τους σε μια ηθική κοινότητα. Στις τροπολογίες 25 και 19 τονίζω ότι πρέπει να έχουμε μια σαφή υποστήριξη προς την Γεωργία. Δεν θέλουμε να διαιωνιστεί η, η σχέση σύνδεσης ως οριστική μορφή των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Γεωργία θέλουμε εν καιρό να οδηγήσουν όλα αυτά στην πλήρη ένταξη της Γεωργίας ώστε η Γεωργία να γίνει πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά τα οποία έχουν επιτευχθεί μετά την Επανάσταση των Ρόδων τώρα βρίσκονται σε κίνδυνο μετά από όλα αυτά που έγιναν σε βάρος των ε, εθνικών κινημάτων και σε βάρος του Πρόεδρου Σακιασβίλη. Αν δεν ασκηθεί πίεση από τον δυτικό χώρο, η Γεωργία και πάλι θα βρεθεί σε πολιτικό αδιέξοδο. Δεν μπορούμε να βασιζόμαστε μονάχα σε αντίπεινα και να δεχόμαστε να ασκούνται αντίπεινα σε βάρος της αντιπολίτευσης στην ε, Γεωργία, αυτό το οποίο βλέπουμε. Θα πρέπει λοιπόν να υπογραμμίσουμε στο ψήφισμά μας και το ρόλο της ε, κοινωνίας των πολιτών και των ε, ηθικών αρχών που θα πρέπει να διέπουν τη λειτουργία της κοινωνίας. Προτείνω λοιπόν να τονίσουμε ιδιαίτερα και το ρόλο της Εκκλησίας. Το ρόλο της Ορθόδοξης Εκκλησίας που παίζει ένα κεφαλαιόδη ρόλο στη χώρα αυτή, γιατί με τον τρόπο αυτό μπορούμε να, να υποστηρίξουμε τη δημιουργία της εθνικής συνείδησης. Θέλω να τονίσω επίσης ότι η ρωσική κατοχή των περιοχών της ε, Γεωργίας είναι μια πραγματική κατοχή. Δεν είναι απόσχηση, δεν είναι περιοχές οι οποίες έχουν αποσκητήσει. Δεν είναι αποτέλεσμα εμφυλίου πολέμου. Αυτά που έγιναν το 2008 έγιναν με την εισβολή του στρατού της Ρωσίας στην περιοχή αυτή και ουσιαστικά έφερε τις περιοχές αυτές στην σφαίρα επιρροή της Ρωσίας. Είναι μια πραγματική λοιπόν εισβολή. Αν θέλουμε λοιπόν να ενισχύσουμε τη γεωργία, να ενισχύσουμε τη σύνδεση της γεωργίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε αυτό το κέριο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η γεωργία. Και αυτό βρίσκεται στην πηγή όλων των άλλων προβλημάτων που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η γεωργία. Και είναι συγκεκριμένα το γεγονός ότι έχουμε την εισβολή αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Αν δεν υπάρχει κάποιος άλλος ο οποίος θα αναλάβει το λόγο, θα ξαναδώσω το λόγο στον κύριο Μανικίνης. Συγγνώμη, υπάρχει κάποιος ακόμα που έχει στήσει το λόγο. Άκουσα τον συνάδελφο Γιούρεκ Έχω παρακολουθήσει τα γεγονότα στη Γεωργία για τον πρόεδρο Σαρκοζή και ε, για τον Γενικό Γραμματέα των Ηλυσίων. Και πράγματι η κατάσταση δεν είναι όλα καλά και όλα άσχημα. Δεν υπάρχουν από τη μία οι κακοί Ρώσοι και από την άλλη οι επαναστάτες της ελευθερίας. Όχι. Έχουμε να κάνουμε με δύο διαφορετικές εξουσίες που επιδιώκουν διαφορετικά συμφέροντα, συμφέροντα που παίζουν ανάμεσα στους Αμερικανούς και τους Ρώσους, ανάμεσα στη Δύση και τους Ρώσους. Ο Γιούρεκ γνωρίζει ότι εγώ ήμουν εταντίος του Σταλινισμού, δεν έχουμε πια το Στάλιν, μας τελείωσε. Ε, πρέπει αγαπητοί συνάδελφοι και αυτή είναι και η άποψη του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να κρατήσουμε το μέτρο και την ισορροπία. Αν αναζητούμε την ειρήνη, αν όμως αναζητούμε την πολιτική σύραξη και αν θέλουμε εμείς ε, να καταδικάζουμε και να αντιπαραθέτουμε το καλό με το κακό και μόνον αυτό, λύσεις στα προβλήματα αυτά δεν θα βρούμε. Λυπάμαι γι' αυτό. Η κυρία Φωτίγκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε κύριε Πρόεδρε. Μετά από αυτά τα οποία άκουσα από τον Γάλλο συνάδελφο, θα ήθελα να, σας, να μου επιτρέψετε να σας υπενθυμίσω το εξής κυρίες και κύριοι ότι το έθνος των ε, Γεωργιανών είναι ένα παλαιό έθνος, είναι ένα έθνος με μεγάλη ιστορία, είναι ένα έθνος παλαιότατο και τα πρώτα μνημεία ε, του Γεωργιανού έθνους ε, πηγαίνουν πίσω στον 5ο αιώνα μετά Χριστόν. Έχουμε πολύ λίγους πολιτισμούς σε αυτό το κομμάτι του κόσμου τόσων παλαιούς. Πρόκειται για μνημεία χριστιανικά, τα οποία κατεστράφησαν συστηματικά και βομβαρδίστηκαν συστηματικά από τις ε, ε, ρωσικές δυνάμεις. Δεν το ξεχνάμε αυτό. όπως θυμόμαστε και τους βομβαρδισμούς κάποιων άλλων σε περιοχές ε, ε, στην, ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο κάποτε πριν από πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, το λέω αυτό γιατί πιστεύω ότι είναι πραγματικά κακό για τη μεγάλη αυτή χώρα, για το μεγάλο αυτό έθνος, να πει κανείς ότι ο αγώνας για την ανεξαρτησία του, ο αγώνας για την αυτονομία του είναι ένα παιχνίδι ε, ανάμεσα σε διαφορετικές συνωμοσίες διεθνούς τύπου. Ο εισηγητής, εν πάση περιπτώσει, έχει το λόγο, λέει ο κ. Μπροκ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις παρατηρήσεις σας, να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που πήραν το λόγο. Βλέπω ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κάποιες ε, συμβιβαστικές λύσεις. Αυτά τα οποία είπαμε όλοι για την επιλεκτική εφαρμογή της δικαιοσύνης είναι κάτι το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και είμαι βέβαιος ότι θα μπορέσουμε ε, να ε, καταλήξουμε σε μια συμβιβαστική πρόταση. Ε, μια διαδικασία η οποία θα είναι ανοιχτή μέχρι την ψηφοφορία τον μήνα Νοέμβριο ε, στην Επιτροπή μας ε, και στην Ολομέλεια αργότερα. Τίποτα άλλο προς το παρόν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σιγητά. Στις 17 Νοέμβρη θα ψηφίσουμε και θα έχουμε προηγουμένως την ευκαιρία να συζητήσουμε για τις τροπολογίες. Η ελπίδα μου είναι ότι ο εισηγητή και οι σκιώδε εισηγητέ θα μπορέσουν να καταλήξουν σε συμφωνία σε σχέση με αυτέ τι τροπολογίε. Και ξέρουμε ότι η Επιτροπή ΙΝΤΑ στις 7 Νοεμβρίου θα καταλήξει σε μια απόφαση σε σχέση με την γνωμοδότηση αυτή, ώστε ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε στην Ολομέλεια του Δεκεμβρίου να υπάρξει η οριστική απόφαση και έτσι να είναι και η χώρα αυτή η οποία η συμφωνία αυτή με τη χώρα αυτή θα μπορέσει η συμφωνία σύνδεση να κυρωθεί. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ισηγητά και ερχόμαστε τώρα στο θέμα της Ουκρανίας. Θα λάβει χώρα μια ανταλλαγή απόψεων με την κυρία Τεσουλουέτα η οποία είναι αρμόδια μαζί με τον κύριο Πλάνκοβα, Πλάνκοβιτς, ο οποίος ήταν ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην ε, Ουκρανία και χαίρομαι πάρα πολύ αν θα μπορούσαν να μας παρουσιάσουν την κατάσταση σε σχέση με τις ούτως υπήν εκλογές που έλαβαν χώρα την Κυριακή στην ε, Ουκρανία. Θα ήθελα λοιπόν να δώσω καταρχήν το λόγο στην κυρία Σουλουέτα, η οποία είναι επικεφαλής της αντιπροσωπείας του ΟΑΣΕ και του Ιδρύματος για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Και στη συνέχεια θα μπορούσε ο κύριος Πλένκοβιτς να μας δώσει και, τη, και στοιχεία από τη δική του πλευρά και φυσικά και οι άλλοι συνάδελφοι που ήταν σε αυτή την αντιπροσωπεία. Κυρία Σουλουέτα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταλαβαίνω γιατί θέλουμε να μιλήσουμε για τις 26 Οκτωβρίου και όχι για αυτά που έγιναν την περασμένη Κυριακή στον Τον Μπάς. Γι' αυτό δεν έχω να πω τίποτα γιατί δεν στείλαμε παρατηρητές εκεί. Το πρώτο που θα ήθελα να κάνω είναι να σας ευχαριστήσω κύριε Πρόεδρε και κύριοι Βουλευτέ για την πρόσκλησή σας. Είναι η τρίτη μου επίσκεψη εδώ και χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό. Κάτι για την παρατήρηση των εκλογών στην Ουκρανία από τον ΟΑΣΕ η αντιπροσωπεία ήταν αρκετά μεγάλη, όχι τόσο μεγάλη όσο για τις προεδρικές εκλογές του Μαΐου, αλλά αποτελούνταν από 700 άτομα. Φτάσαμε στην Ουκρανία στις 7 Οκτωβρίου, στις 27 Οκτωβρίου αναπτυχθήκαμε όλοι και τελειώσαμε την αποστολή την Παρασκευή αυτή την εβδομάδα. Εκείνη την εβδομάδα δηλαδή δεν παρατηρήσαμε τίποτα, δεν στείλαμε παρατηρητές στις αποσχιστικές περιφέρειες που θέλουν την ένωση με τη Ρωσία. 27 λοιπόν από τις νέες έδρες στην Ουκρανία θα παραμείνουν κενές γιατί έπρεπε να προέρχονται από εκείνες τις περιφέρειες. 39 χώρες συν την Ιαπωνία έστειλαν παρατηρητές 18 από τη Ρωσική Ομοσπονδία. 90 παρατηρητές χρηματοδοτήθηκαν από την Ένωση. Μπορέσαμε να συντονίσουμε όλες μας τις προσπάθειες την ημέρα, την ημέρα των εκλογών όπου είδαμε περίπου 200 κοινοβουλευτικούς παρατηρητάς και ήρθαν επίσης και από από τον Άτο, από τον ΟΑΣΕ και τα λοιπά. Και επιβλέψαμε περίπου 3.000 εκλογικά τμήματα. Συμπληρώθηκαν χαρτιά 4.000 περίπου και όπως ξέρετε η αποτίμησή μας ήταν γενικά θετική ιδιαίτερα για την ημέρα των εκλογών όπου τα πράγματα ήταν καλά οργανωμένα με εφταξία και 99% από τα εκλογικά τμήματα δεν αντιμετώπισαν κανένα διαδικαστικό πρόβλημα. Αυτό συμφωνεί με τις παρατηρήσεις που κάναμε σε όλα τα εκλογικά τμήματα και τις περιφέρειες. Βέβαια, επαναλαμβάνω, δεν στείλαμε κανέναν στον Ντονέτσκ και τον Λουγκάνσκ Μόνο στο Σλαβιάνσκ στείλαμε μερικούς εκπροσώπους. Όπως και στις προεδρικές εκλογές της Άνοιξης παρατηρήσαμε ότι η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή που οργάνωσε τα πράγματα τα έκανε πολύ καλά και αυτή τη φορά. Τηρήθηκαν όλα τα χρονοδιαγράμματα και με πολύ αποτελεσματικό τρόπο. Παρατηρήσαμε και μερικές δυσκολίες που αφορούν όμως ακριβώς το ότι ήρθαν πάρα πολύ προσήλθαν πάρα πολλοί να ψηφίσουν. Και συγχαρήκαμε τους ε, πολίτες της Ουκρανίας για τον φιλήσυχο τρόπο με τον οποίο ε, διέπραξαν, έπραξαν αυτά του τα εκλογικά καθήκοντα. στις δύο περιφέρειες Λουχάνσκ και Ντονέτσκ που ελέγχονται από τους αποσχιστικούς δεν υπήρξαν προβλήματα ούτε εκεί παρά το ότι συνεχίζονται οι διαμάχες και, σειράξεις συγκρούσεις. Στην, την ημέρα των εκλογών σημειώθηκαν δύο νέα κρούσματα και την τελευταία εβδομάδα το σύνολο έφτασε τα 21. Η αποστολή μας επίσης σημείωσε ορισμένα μεμονωμένα βία, ορισμένες βίες, βιοπραγίες. Δεν είχαμε κάνει τελείως θετική αποτίμηση για όλες τις περιεκλογικές περιφέρειες γιατί 19 περιφέρειες, σε 19 περιφέρειες Σημειώθηκαν βιοπραγίες εξών 16 στις αποσχιστικές περιοχές. Πρέπει να σημειωθεί ότι σε μερικές περιφέρειες όπως ο Λουχάν και το Ντονέσκ περιορίστηκαν οι εκλογές σε μόνο λίγα εκλογικά τμήματα όπως στο Λουχάνκ 4. Γενικά όμως τονίζω όπου υπήρξαν προβλήματα οφείλονται στον υψηλό αριθμό των προσερχομένων εκλογέων δεν παρατηρήσαμε καμία κακή χρήση των διατεθειμένων πόρων, πράγμα που στο παρελθόν ήταν πρόβλημα, αλλά ο πρόεδρος και πρωθυπουργός απευθύνθηκαν στην τηλεόραση καταχρηστικά, γιατί δεν θα έπρεπε την ημέρα των εκλογών να γίνουν πολιτικές δηλώσεις. Στείλαμε παρατηρητές και σε έξι εθνικά και δύο ιδιωτικά τηλεοπτικά δίκτυα και μπορώ να πω ότι υπάρχει πολύ μικρή ανεξάρτητη ειδησιογραφία αλλά έγιναν προσπάθειες από τη δημόσια τηλεόραση για μια πιο αντικειμενική ενημέρωση. το ειδικό όργανο για την ε, διασφάλιση της αντικειμενικότητας της ενημέρωσης πάντως ίσως να αντιμετώπισε μπορούμε να πούμε ορισμένες ελλείψεις. Από τα 29 κόμματα που κατέβηκαν τις εκλογές μόνον 6 εξέλεξαν ε, εκπροσώπους. Το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι εκτός Βουλής και η κατανομή των εδρών με βάση τουλάχιστον το 99,9% της καταμέτρησης είναι ότι ο κύριος Ποροσένκο, το κόμμα ή συνασπισμός του κύριου Ποροσένκο, 132 έδρες και του Πρωθυπουργού, το λαϊκό μέτωπο του Πρωθυπουργού, 82 έδρες. Η εκπλήξη είναι το κόμμα αυτοδιάθεση που έχει 35 έδρες. Και όπως ξέρετε τώρα γίνονται συνεννοήσεις για συνασπισμούς. Επίσης η αναλογικότητα της προσώπησης των γυναικών είναι απογοητευτική. 47 γυναίκες θα μπουν στο κοινοβούλιο έναντι 43 του προηγουμένου. Είναι πολύ κακή η εκπροσώπηση των γυναικών λοιπόν στις μονοεδρικές περιφέρειες. Τελικά κύριε Πρόεδρε όλοι μας οι συνομιλητές συμφώνησαν ότι έγιναν πολύ καλά οι εκλογές οργανώθηκαν χωρίς ειδικά προβλήματα. Και γι' αυτό θα έπρεπε να σημειώσουμε ότι παρά από ορισμένες διαμαρτυρίες Γενικά κανένα από τα κυριότερα κόμματα δεν αμφισβήτησε τα αποτελέσματα. Επίσης, μας είπαν ότι υπάρχει πολιτική θέληση να ακολουθηθούν οι συστάσεις της ΟΑΣΕ, πρώτη από τις οποίες είναι η έγκριση ενός συνεπούς εκλογικού νόμου. Το θέμα τώρα της χρηματοδότησης των προεκλογικών εκστρατιών δεν έχει αντιμετωπιστεί μέχρι τώρα και σε συνεργασία με τον ΟΑΣΕ και τις αρχές της Ουκρανίας θα προχωρήσουμε στη λήψη νέων μέτρων και προτάσεων στην πρώτη φάση. Απαιτούνται νέοι κανόνες για την μεγαλύτερη σταθεροποίηση της διαχείρισης των εκλογών, ιδιαίτερα για τους καταμετρητές ψήφων. Ελπίζω λοιπόν ότι μετά από τη θετική ανταπόκριση ε, την οποία δείξατε απέναντι ε, στην αποστολή μας αυτή θα μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε μια μονιμότερη επαφή με τις αρχές της Ουκρανίας που θα οδηγήσει πιο εύκολα στις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται στο εκλογικό σύστημα. Σας ευχαριστώ, εισηγητής, κύριος Πλένκοβιτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ξεκινώντας θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που είναι μέλη της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την Ουκρανία και είναι παρόντες σήμερα εδώ. Θα ήθελα να καλωσορίσω επίσης και τα μέλη της, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πήραν μέρος στις πρόορες εκλογές που διεξήχθησαν στην Ουκρανία. Να ευχαριστήσω επίσης και την κυρία Ζουλουέτα και γενικά όλους τους εκπροσώπους και της, ε, ε, της ε, υπηρεσίας εξωτερικών σχέσεων διότι κάλυψαν με λεπτομέρεια και επιμονή και το νομικό πλαίσιο, το εκλογικό πλαίσιο και την κάλυψη των προεκλογικών διαδικασιών από τα μέσα ενημέρωσης και τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας και την αξιολόγηση στο τέλος. Υπάρχουν δύο θέματα τα οποία καλούμεθα να συζητήσουμε σήμερα για τις πρόορες αυτές εκλογές. Το ένα θέμα είναι οι διαδικασίες. Εδώ νομίζω ότι η κυρία Ντεσουλουέτα πάρα πολύ ε, σωστά είπε ότι η νέα ράντα της Ουκρανίας έχει αυτή τη στιγμή 450 βουλευτές 225 ε, σε συγκεκριμένες εθνικές, ε, ε, εθνικούς καταλόγους, αλλά δεν θα καλυφθούν όλες οι θέσεις όπως προβλέπει το, Σύνταγμα, γιατί 27 βουλευτές από την Κρυμαία, 9 από τον Ντόνετς και 6 από το Λουχάνσκ δεν μπόρεσαν να εκλεγούν και θα υπάρχουν λιγότερες θέσεις χειρεύουσες πλέον αλλά ταυτόχρονα σύμφωνα και με το Ουκρανικό σύστημα, σύνταγμα, συγγνώμη, απαιτείται ε, κατελάχιστον η εκλογή 350 βουλευτών για να θεωρηθεί έγκυρη εκλογή και στη συγκεκριμένη περίπτωση κάτι τέτοιο ισχύει. Λοιπόν, εγώ μπορώ να σας μεταφέρω τις εντυπώσεις των Ευρωβουλευτών που πήγαν εκεί. Ε, οι εκλογές διεξήχθησαν με τακτικό τρόπο, με σωστό τρόπο. Πήγαμε και στο Κίεβο, στο Χαρκίβ, στην Οδυσσό, στο Τσερκάσκι και στο Δινοπετρόσκ. Οι πληροφορίες τις οποίες συλλέξαμε από τους συναδέλφους που ε, ήσαν εκεί είναι ότι οι εκλογές εξελίχθησαν καλά με ειρηνικό τρόπο και όλοι οι συνάδελφοι είδαν ότι δεν υπήρχαν σημαντικές δυσκολίες. Βρισκόμαστε λοιπόν στα πλαίσια της διαδικασίας διατύπωσης των προκαταρτικών ευρημάτων σε συνεργασία με τις αντιπροσωπείες του ΟΑΣΕ, του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Κοινοβουλευτικής Συνελεύσεως του Βορειοατλαντικού Συμφώνου. Νομίζω ότι ε, έχουμε καλύψει ένα μεγάλο έδαφος, αλλά και οι συνάδελφοι αυτοί έχουν καλύψει ένα ευρύτερο, μια ευρύτερη γεωγραφική περιφέρεια και συλλέγουμε όλα τα στοιχεία, ακόμα και τις επιμέρους κριτικές, οι οποίες συνιστούν ένα επιπλέον κίνητρο για την Ουκρανική κυβέρνηση για να κάνει τις αλλαγές οι οποίες ε, απαιτούνται. Υπήρξε πρόοδο σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές και τις προεδρικές εκλογές και θα υπάρξει πρόοδος ελπίζω και στις επόμενες οι οποίες θα οργανωθούν σύμφωνα με τα διεθνώς αναγνωρισμένα επίπεδα η συμμετοχή ήταν πάνω του 50%, χαμηλότερη του αναμενωμένου πάντως, παρόλα αυτά ήταν μια αρκετά ισχυρή συμμετοχή αν συγκρίνουμε ε, με το τι συμβαίνει στις δικές μας κυρίως χώρες. Ε, θα πρέπει επίσης να σημειώσουμε, και αυτό έχει μεγάλη σημασία, είναι ότι οι εκλογές της 26 Οκτωβρίου αποτελούν τμήμα μιας ε, διαδικασίας σε τρία στάδια μετά από το Ευρωμαϊντάν, μετά από τις προεδρικές εκλογές τον Μάιο, αυτή η ευκαιρία την οποία διείδε ο πρόεδρος Πόροσένκο για τις πρόορες εκλογές για να υπάρξει μια νέα αναγνωρισμένη πλέον ράντα μας ε, οδήγησε σε ένα νέο πολιτικό τοπίο πλέον και τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η πλειοψηφία των Ουκρανών επιλέγουν την Ευρώπη, επιλέγουν τις μεταρρυθμίσεις, επιλέγουν όμως και την ενότητα και την εδαφική ακαιρεότητα της χώρας τους. Ως εκ τούτου εδώ ε, διακρίνουμε τη μεγάλη σημασία που έχει και η διαδικασία και συμφωνία του Μίνσκ όπως επίσης ε, και η Συμφωνία των Βρυξελών για την αναβολή της Συμφωνίας της Εταιρικής μέχρι το 2016 και σημειώνουμε και την πρόοδο που συνετελέστη για τις, στις διαπραγματεύσεις ε, των Υπουργών Ενέργειας ε, για το θέμα της προμήθειας φυσικού αερίου. Όλα αυτά τα στοιχεία δημιουργούν μια κατάσταση πιο ειρηνική θα έλεγα από ό,τι στο παρελθόν. Ε, ανάμεσα στις δύο προηγούμενες εκλογές 3.500 ε, κόσμος και πάνω από 3.500 κόσμος ε, έχασε τη ζωή του. Πολλά τμήματα της χώρας αυτής είχαν αποκλειστεί και είδαμε ιδιαίτερα στις συναντήσεις που είχαμε με τους Ποροσένκο, Γιατσένιοκ και Τουρτσίνοφ, τον πρόεδρο της Νέας Ράντα, όπως επίσης και τον προηγούμενο υποψήφιο πρόεδρο Κλίντσικ, ότι έχει υπάρξει σημαντική πρόοδος όπως και ε, ε, υπάρχει πάντα ο στόχος βέβαια της επανένωσης με ειρηνικό τρόπο του συνόλου της Ουκρανικής επικράτειας. Υπάρχουν πολλές προσδοκίες από πλευράς των Ουκρανών φίλων για τη συμφωνία και νομίζω ότι η υποστήριξη η οποία απεδείχθη από πλευράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλων ευρωπαϊκών οργάνων ε, προς τους Ουκρανούς είναι σημαντική παρακαταθήκη για το μέλλον της χώρας. Τώρα για τις χθεσινές εκλογές. Όλοι μας ε, νομίζω θεωρούμε ότι είναι παράνομες, ε, αθέμητες και αντίθετες με την Ουκρανική νομοθεσία. Δεν θα αναγνωριστούν τα αποτελέσματα αυτά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και κάθε προσπάθεια της Μόσχας να τις νομιμοποιήσει είναι κατά της συμφωνίας του Μίνσκ και υπονομεύει τις προσπάθειες επίτευξης ειρηνικής λύσης. Στο τέλος λοιπόν αυτών των σύντομων σχολείων, γιατί όπως σας είπα η γραπτή έκθεση των αποτελεσμάτων της εκλογικής παρατήρησης θα κυκλοφορήσει σε λίγες εβδομάδες. Θέλω να ευχαριστήσω απλά στην παρούσα φάση τους συναδέλφους, τον Αντιπρόεδρο, τον κύριο Τσαρνέσκι, την κυρία Κοράτσα Μπίλκ, Τσούρεκ, Ντέμερ Σμάκε, Βαν Μπάλεν, Αυστρεβίτσιους, Ράνσδορφ, Χάρμς και όλους τους συναδέλφους για την συνεργασία τους στην αποστολή την οποία αναλάβαμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συμφωνήσω με αυτά που είπε ο κύριος Πλένκοβιτς προηγουμένως. Δύο ίσονες παρατηρήσεις τώρα, αν μου επιτρέπετε, για να προσθέσω σε αυτά που είπε ήδη ο κύριος Πλένκοβιτς. Πρώτα απ' όλα, Χρειαζόμαστε να εκφράσουμε με πιο στεντόρια φωνή τη θέση μας ότι η, ευρωπαϊκή προσέγγιση σημαίνει μεγαλύτερη παρουσία γυναικών σε ένα κοινοβούλιο όπως το Ουκρανικό Κοινοβούλιο. Δεύτερον, θα πρέπει να συγχαρούμε με ένα έκτακτο τρόπο, με ένα ιδιαίτερο τρόπο την διεξαγωγή των εκλογών στην Ουκρανία γιατί ήταν πάρα πολύ δύσκολο το εγχείρημα αυτό. Φανταστείτε τώρα μια χώρα που σε πολλές περιοχές είναι εμπόλεμες ουσιαστικά συνθήκες όπου υπάρχουν πολλές διεθνείς εντάσεις στη χώρα αυτή το ότι μπόρεσαν με ο τρόπο ομαλό και θετικό να διοργανώσουν την παρουσία 900 ξένων παρατηρητών για τις εκλογές, κάτι το οποίο θα μπορούσε να ήταν ένα μεγάλο άχθος για τους οργανωτές. Το γεγονός ότι είναι με επιτυχή τρόπο, με επαγγελματικό τρόπο, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θέλουμε να συγχαρούμε λοιπόν τους Ουκρανούς για αυτό. Και μια τελευταία παρατήρηση Θέλουμε να συγχαρούμε φυσικά και τον κύριο Πλένκοβιτς για, το δικό του ρόλο στην παρακολούθηση των εκλογών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα μιλήσω, στα Ολλανδικά που είναι η μητρική μου γλώσσα. Θέλω και εγώ να συγχαρώ, να ευχαριστήσω τον κύριο Πλένκοβιτς και όλους τους συναδέλφους για την εξαιρετική μας συνεργασία κατά την αποστολή στην Ουκρανία. Πράγματι εκεί ζήσαμε αληθινές και σωστές εκλογές, έγιναν σεβαστές όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες και αποτέλεσμα ήταν τώρα να υπάρχει μια σωστή εκπροσώπηση του λαού, αληθινή εκπροσώπηση του λαού μετά την φυγή του Γιαννουκόβιτς και τα γεγονότα στο Μαϊντάν. Και τώρα μπορεί το Κοινοβούλιο να εφαρμόσει μεταρρυθμίσεις εν πλήρη νομιμότητη. Μπορεί κανείς λοιπόν πια να μιλήσει όντως για πλειοψηφία η οποία θέλει μεταρρυθμίσεις και θέλει μια σύγχρονη και μοντέρνα δημοκρατική κοινωνία. Εγώ πήγα και στην Οδυσσό όπου όλα έγιναν επίσης ειρηνικά αλλά αλλά λέγω δεν υπήρξε εκλογική συμμετοχή των εσωτερικών προσφύγων που είναι πάρα πολλοί από τον Ντονμπάς. Αυτοί δεν συμμετέσχουν στις εκλογές παρά το ότι οι αρχές είχαν διευκολύνει την εγγραφή τους στους εκλογικούς καταλόγους, δεν τους παρεμπόδισαν. Και ερωτώ, οι αρχές λοιπόν Μήπως δεν τους κινητοποίησαν αρκετά, μήπως δεν τους ευαισθητοποίησαν αρκετά. Γιατί στις ανατολικές επαρχίες, από τις ανατολικές επαρχίες υπάρχουν 400.000 εσωτερικοί πρόσφυγες και αυτοί δεν συμμετέσχουν καθόλου στις εκλογές αυτές και άρα δεν εκπροσωπούνται στη Βουλή. Και οι νέοι διαπίστωσα ότι προσήλθαν πολύ λίγοι νέοι στις εκλογές. Υπάρχει βέβαια το διπλό εκλογικό σύστημα που συνήθως το συνδυάζουμε με την εκλογική διαφθορά. Αλλά για την απουσία των νέων δεν καταλαβαίνουμε. Ίσως υπάρχει απλώς λιγότερη εμπιστοσύνη. Ελπίζω μετά τη μεταρρύθμιση του εκλογικού νόμου να υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή των νέων. Γιατί πρέπει πρωτίστως να αλλάξει ο εκλογικός νόμος. Γιατί όταν βλέπουμε τι γίνεται στον Ντονμπάς και στις ανατολικές επαρχίες γενικότερα, είδαμε εκεί τις ψευτοεκλογές, αλλά τοπικά, τοπικά, μήπως χρησιμοποιηθούν από τους Ρώσους αυτοί οι άνθρωποι για να νομιμοποιηθούν οι παρανομίες των μήπως θελήσουν οι Ρώσοι να αρπάξουν και άλλες περιοχές. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει αφοπλισμός τους και μεγάλη πίεση επί της Ρωσίας ως προς αυτό. Τέλος. Εκτός από τις ίδιες μου τις εμπειρίες στην Οδύσσο, άκουσα και νέα από τον Ντονέτσκ και φαίνεται ότι εκεί πίεζαν τον κόσμο κάτι ιδιωτική στράτη που πίεζαν τον κόσμο για να ψηφίσει όπως τους έλεγαν αυτοί. Τώρα, κατά πόσον αυτή η επιρροή επηρέασε και το τελικό αποτέλεσμα, δεν ξέρω, εγώ απλώς κάτι νέα άκουσα. Ευχαριστώ κύριε Ζάμσταφ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήμουν κάπως πιο σκεπτικιστής από ορισμένους συναδέλφους. Εγώ ήμουν στην περιοχή του Νιεφροπετρόφσκ που είναι ήταν μία από τις περιοχές όπου έγινε η παρακολούθηση. Εκεί μπορώ να πω ότι υπήρξαν κάποιες παραβιάσεις του εκλογικού νόμου. Καταρχήν υπήρξε τρομοκράτηση των ε, ψηφοφόρων από την συνεχή παρουσία ατόμων που ήταν ε, με στρατιωτικές στολές και ένοπλοι στα εκλογικά τμήματα. Αυτό δεν είναι ακριβώς κάτι το οποίο θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι συνάδει με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, αλλά συνέβη πολλές φορές. Επίσης υπήρχαν πληροφορίες για αγορά ψήφων με μέσο κινητού τηλεφώνου και επίσης υπήρξαν και άλλες λαθροχειρίες γιατί παραδείγματος χάρη τα αποτελέσματα των, της ψηφοφορίας σε κάθε εκλογικό τμήμα απεστάλησαν στα κεντρικά γραφεία, αλλά από εκεί αναμεταδόθηκαν με μια παραποιημένη μορφή. Αυτό δεν έγινε μονάχα μια φορά, το είδα σε διάφορες περιπτώσεις να λαμβάνει <clears throat> χώρα. Εγώ χρησιμοποίησα τους ε, συνεργάτες μου και δημιούργησα δίκτυα πληροφόρησης στην περιοχή αυτή. Έχω λοιπόν πολλές ε, περιπτώσεις που μπορώ να αναφέρω σε, αυτές τις, σε ό,τι αφορά λαθοχειρίες. Επίσης υπήρξε βία που χρησιμοποιήθηκε πριν από τις εκλογές και κατά τη διάρκεια των εκλογών στους δρόμους των περιοχών αυτών. Και υπήρξε και μια <clears throat> χρήση βίας και τρομοκράτησης εναντίον του Κομμουνιστικού Κόμματος και των κομμάτων της αντιπολιτευσής. Υπήρξε καταστροφή εκλογικού υλικού ορισμένων κομμάτων όπως του Βατκευσίνα και άλλων. Πρέπει να σας πω λοιπόν ότι θα πρέπει να παρακολουθήσουμε προσεκτικά και στο μέλλον την κατάσταση στην Ουκρανία. Υπήρξε κατά την άποψη των ε, παρατηρητών ότι υπήρχε κίνδυνος να μην κερδίσουν οι ευρωπαϊκά οι προσκύμενες προς την Ευρώπη δυνάμεις και τότε αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μην ανοίξουν καν τα εκλογικά τμήματα σε αυτή την περιοχή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ και τους δύο πρόεδρους των αντιπροσωπιών παρατήρησης των εκλογών της Ουκρανίας, την κυρία ε, Θουλουέτα και τον κύριο Πλένκοβιτς να τους ευχαριστήσω και όλους τους συναδελφούς που πήγαν εκεί. Είχα κάποιες σύντομες ερωτήσεις να θέσω για τους ε, μακροπρόθεσμους και τους βραχυπρόθεσμους παρατηρητές, αν μπορούν να μας πούν πόσοι ε, ρωσόφωνοι συμμετέσχαν στις εκλογές. Και επίσης πώς θεωρείτε ότι θα αντιμετωπίσει η Ρωσία ως μέλος της ΟΑΣΕ τα συμπεράσματα από την παρακολούθηση των εκλογών. Δεύτερον, πρέπει να πω ότι το εκλογικό σύστημα το οποίο χρησιμοποιήθηκε δεν είναι το καλύτερο για μια χώρα η οποία προχωρά προς τη δημοκρατικοποίηση ε, και δεν συνάδει με τις ε, συστάσεις της Επιτροπής της Βενετίας του Συμβουλίου της Ευρώπης. Θα ήθελα να ξέρω λοιπόν αν υπάρχει η θέληση να ληφθούν υπόψη αυτές οι προτάσεις της Επιτροπής της Βενετίας για τις μεταγενέστερες εκλογές και αν θα υιοθετηθούν. Ευχαριστώ. Ο πρώτος χωρίς μικρόφωνο αναφέρει το όνομα του επομένου μιλητή που είναι η κυρία Γκόμες. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δύο επικεφαλής αντιπροσωπείας. Θα ήθελα να ενθαρρύνω η έκθεση να είναι λεπτομερής να περιλαμβάνει και τα σημεία κριτικής, τις ελλείψεις και τις απαιτούμενες και απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Γνωρίζουμε το τι θέλουμε να γίνει στην Ουκρανία, αλλά η αποκατάσταση της δημοκρατίας απαιτεί, θα έλεγα, πάρα πολλές ε, ε, μεταρρυθμίσεις. Μπορούμε λοιπόν να είμαστε πολύ πιο συγκεκριμένοι στις ε, ε, παρατηρήσεις και τις προτάσεις τις οποίες θα κάνουμε. Πάρα πολύ λίγοι νέοι Ουκρανοί πήραν μέρος στις εκλογές και αυτό είναι κάτι το οποίο μας ε, απασχολεί ιδιαίτερα. Και αυτό αποδεικνύει την ανάγκη για πραγματικές μεταρρυθμίσεις. Μια ανάγκη η οποία φυσικά αισθάνονται πρώτοι οι πολίτες της χώρας. Σας ευχαριστούμε πάντως Πρόεδρε που αναφερθήκατε και μέσω της δηλώσεώς σας στο θέμα της νομιμότητας των λεγόμενων εκλογών του Ντονμπάς. Πάντα η δημοκρατία και οι προτάσεις οι οποίες έγιναν προς τους λαούς της περιοχές είναι κάτι το οποίο φυσικά δημιουργεί προβλήματα και αυτά το οποίο συνέβη χθε δεν ήταν εκλογές πολύ απλά. Και στο Χάρκοβο, στο Χαρκίβ, θα ήθελα να πω, λέει ο κύριος Φανμπάλεν, ο κόσμος ε, ε, ψήφισε ειρηνικά. Δεν δημιουργήθηκαν προβλήματα για μένα και για την ομάδα στην οποία ήμουν μέλος. Δεν υπήρξαν προβλήματα γενικά και αναφέρομαι σε μια περιοχή η οποία είναι κυρίαρχα ρωσόφωνη. Αυτή ήταν η εικόνα την οποία εν πάση εμείς σχηματίσαμε. Θα συμφωνήσω με την κυρία Γκόμες ότι οι εκλογές στην περιοχή Ντόνμπας είναι κάτι το απαράδεκτο και είναι μια προφανής παραβίαση της συμφωνίας του Μίνσκ. Τώρα, ε, πρέπει να συνεργαστούμε σωστά με τους Ουκρανούς φίλους και να πω επίσης ότι η λεγόμενη φασιστική άκρα δεξιά, την οποία αναφέρει συνεχώς η Μόσχα, δεν την είδαμε πουθενά και δεν εξελέγησαν οι άνθρωποι αυτοί πουθενά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία αυτή που έχουμε να ανταλλάξουμε, να ανταλλάξουμε απόψη για το θέμα αυτό. Διάβασα προσεκτικά τις εκθέσεις. Εγώ τώρα θα πρέπει να διαφωνήσω. Είναι άχαρο το έργο μου. Θα πρέπει να θυμηθούμε όλοι τι υπήρξε προηγουμένως. Ότι υπήρξε μία κατάσταση ανατροπής μιας κυβέρνησης που οδήγησε σε ενόπλες συνθήκες υπάρχουν εξωτερικοί παράγοντες που δεν θέλουν να υπάρξει μια πραγματική ευρωπαϊκή πολιτική καλής γειτονίας. Για τις εκλογές τώρα πώς έλαβαν χώρα. Δείχνουν ότι είναι μικρή τα στοιχεία, ότι είναι μικρή η συμμετοχή, λίγη περιορισμένη η υποστήριξη <clears throat> στην κυβέρνηση και λιγότερο από 30% των δυνάμεων που υποστηρίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω λοιπόν ότι οι εκλογές που δεν οδηγούν σε μια καλύτερη κοινωνική συνένεση δεν μπορούν να βοηθήσουν μια κοινωνία να προχωρήσει. Δεν μου αρέσει λοιπόν το να μιλάτε συνέχεια για τη Ρωσία που να είναι πάντα ε, υπεύθυνη. Μου θυμίζουν αυτά που έλεγε ο Σεράνο Σούνιερ την εποχή του Φράνκο. Πολλές φορές υπάρχει συνεργασία και για την, από τη ρωσική πλευρά για την Ουκρανία σε αυτά που γίνεται. Γι' αυτό θέλω να τονίσω ότι είναι σημαντικό να υποστηρίξουμε την καλύτερη συνένεση μέσα στην Ουκρανία, τη συμμετοχή όλων των δυνάμεων για να οργανωθεί καλύτερα το κράτος και η κοινωνία και μόνο έτσι μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτές τις ε, διαφορές. Κύριε Σαφχάουζερ, ήσασταν και εσείς παρών την Κυριακή στις παράνομες εκλογές στο Ντονμπάς, ίσως μπορείτε να μας δώσετε και κάποια στοιχεία σε σχέση με τα κόμματα τα οποία έλαβαν χώρα σε αυτές τις εκλογές ώστε να έχουν επιλογή οι πολίτες εκεί. Ίσως μπορείτε να μας πληροφορήσετε καλύτερα για τα θέματα αυτά. Είναι πολύ ενδιαφέρον να ξέρουμε για κάποιον <clears throat> ο οποίος προέρχεται ε, από τη Γαλλία μπορεί να αντιμετωπίσει το θέμα της ε, λειτουργίας των εκλογών που συμμετέσχαν πολλές σταλινικές δυνάμεις εκεί. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήμουνα στο Ντομπάς και γύρισα μόνο πριν από μερικές ώρες εδώ στις Βρυξέλλες. Να σας πω καταρχήν ότι θεωρώ ότι οι εκλογές που έλαβαν χώρα την προηγούμενη εβδομάδα, δεν λέω για αυτές που έγιναν την Κυριακή μονάχα. Αυτό ήταν μια απαραίτητη διαδικασία, όπως αναφέρθηκε και από τον συναδελφό μου. Εμείς βρεθήκαμε σε μια κατάσταση όπου είχε υπάρξει μια ανατροπή, ορισμένοι μιλάνε και για πραξικόπημα, θα έπρεπε να μπορέσει να υπάρξει μια νέα κυβέρνηση η οποία να βασίζεται στην εκλογική νομιμοποίηση. Αυτή η διαδικασία λοιπόν ήταν απόλυτα απαραίτητη ακόμα και αν μπορεί να έχουν μια διαφορετική άποψη, όταν ορισμένοι δίνουν ήδη τα, δίνανε ήδη πριν από ένα μήνα τα αποτελέσματα των εκλογών πρωτού λάβουν χώρα αυτέ οι εκλογέ. Δεν θέλω όμω να αναφερθώ σε αυτό το σημείο. Θέλω να πω ότι η κυβέρνηση του Κιέβου επεζήτησε την νομοποίηση από τους ψηφοφόρους στο ανατολικό κομμάτι της Ουκρανίας, όμως έχουμε μια δραματική κατάσταση. <clears throat> Δεν πρόκειται να επισέλθω στις λεπτομέρειες εδώ. Εν πάση υπήρξε βομβαρδισμός του άμαχου πληθυσμού, είδα σχολεία να έχουν βομβαρδιστεί, μου είπανε πάνω από 100 σχολεία, εγώ βέβαια δεν είχα δει τόσα πολλά, είδα νοσοκομεία τα οποία έτυχαν επιθέσεως, είδα τη θέληση να εκδιωχθεί ο πληθυσμός από τις περιοχές αυτές. Μιλάνε για 750.000 άτομα τα οποία εκδιώχθηκαν και μου λένε οι φίλοι μου από την ΟΑΣΕ ότι ο αριθμός των νεκρών είναι της τάξης των 10.000 και όχι πολύ λιγότερο όπως λένε ορισμένοι. Έχουμε λοιπόν ενώπιό μας ένα πληθυσμό με τους οποίους μπόρεσα εγώ να μιλήσω, ένα ενός πληθυσμού ο οποίος είναι τραυματισμένος από όλα αυτά τα οποία έλαβαν χώρα. Είναι γεγονός ότι αυτός ο πληθυσμός, ο οποίος <clears throat> είναι στο μεγαλύτερο βαθμό ρωσόφωνος, δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής τουλάχιστον να αναγνωριστεί η ταυτότητά του. Εγώ δεν είδα να υπάρχει κανένα είδος μίσους που εξεφράστηκε από αυτούς. Τους ρώτησα, μισείτε τους αδελφούς σας που σας βομβάρδισαν. Μου είπαν όχι. Αυτοί που φταίνε είναι οι πολιτικοί. Πληρώνουμε την ύφη μιας σύγκρουσης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας. Έτσι μου είπαν. Βέβαια, όταν έχουμε ένα πόλεμο πρέπει να ξαναβρούμε το δρόμο της ειρήνης. Και για να βρούμε το δρόμο της ειρήνης για μένα υπάρχει μόνο μία λύση, ένας δρόμος έχουμε και στην Ανατολική Ουκρανία μια αυτοανακηρυγμένη εξουσία, η οποία αναζητεί και αυτή μια νομιμοποίηση, γιατί καταρχήν δεν είχε. Και η εκλογική διαδικασία τους επέτρεψε, καλός κακός, αλλά μου λένε οι περισσότεροι περίπου στο ίδιο επίπεδο ε, νομιμοποίησης, όπως και οι εκλογές που έγιναν στο Κίεβο. Τους επέτρεψε να βρουν μια μορφή λοιπόν νομιμοποίησης μέσω των εκλογών. Δεν θεωρώ λοιπόν ότι είναι λογικό να μην αναγνωρίσουμε την εξουσία γιατί κάποια μέρα θα πρέπει να κάτσουμε σε ένα τραπέζι και να συζητήσουμε μαζί του. Θα πρέπει να βρούμε λύσεις για το μέλλον. Θα πρέπει να σταματήσουμε να δαιμονοποιούμε οι μεν τους δε. Θέλουμε να συνεχίσουμε να επιζητούμε τον πόλεμο, να επιζητούμε τη σφαγή των πληθυσμών. Μου είπανε ότι ήρθανε χιλιάδες φορτηγά από τη Ρωσία που ήρθαν στην Ανατολική ε, Ουκρανία. Εγώ στους δρόμους δεν είδα ούτε ένα τέτοιο φορτηγό. Εν πάση περιπτώσει εγώ πήγα, ήρθα, έκανα για τρεις μέρες πολλές διαδρομές, δεν είδα ούτε ένα τέτοιο φορτηγό να έρχεται από τη Ρωσία. Αυτό που σας ζητώ είναι ας προσπαθήσουμε να βρούμε τις βάσεις για ένα διάλογο. Είναι φανερό ότι αυτοί οι πληθυσμοί θέλουν το δικό τους κράτος. Εγώ δεν πήγα εξ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και εκεί ήμουν σαφής. Τους είπα ότι η λύση πρέπει να είναι να βρείτε βάση διαλόγου, να ξαναβρείτε την ενότητα της χώρας σας. Εμείς όμως πρέπει να συμβάλλουμε με το να μην δαιμονοποιούμε τη μία πλευρά ή την άλλη. Δεν νομίζω λοιπόν ότι αγαπητοί συνάδελφοι μπορούμε να προχωρήσουμε. Όλα αυτά που σας λέω λοιπόν θα πιστεύω ότι πρέπει να γίνουν σε λογικό επίπεδο και να δίνουν την εικόνα ενός κοινοβουλίου που επιζητεί την ειρήνη και την ομαλότητα. Ευχαριστώ λέει και ο Πρόεδρος. Η κυρία Καλνιέτε. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τους Ουκρανούς για τις επιτυχείς εκλογικές διαδικασίες. Ευχαριστώ τους συναδέλφους ε, που πήραν το λόγο και μας παρουσίασαν τις εκλογές αυτές, την κυρία Ζολουέτα και τον ε, εισηγητή μας, τον κύριο Πλένκοβιτς. Οι φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις είναι υπεύθυνε τώρα για τις εξελίξεις στη χώρα και τις μεταρρυθμίσεις. Είναι πράγματι μια καταπληκτική ευκαιρία για την χώρα αυτή. Θέλω να ευχαριστήσω και εσάς όμως κύριε Πρόεδρε, όπως και τον κύριο Πλένκοβιτς, για τις ξεκάθαρες θέσεις σας για τις εκλογές στον Τόνμπας. Είναι παράνομες, μη νομιμοποιήσιμες και θα ήθελα να πω στον προηγούμενο μιλητή που επισκέφθηκε τον Ντόνμπας και ο οποίος αναφέρεται πάντα υπέρ του διαλόγου και τα λοιπά που είναι αναγκαιότητα για τις δύο πλευρές, ο διάλογος έχει προταθεί από τις Ουκρανικές αρχές επανειλημμένα και στη Γενέβη και στο Μίνσκ ε, με τη συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός. Αλλά νομίζω ότι οι ε, εκλογές αυτές παραβιάζουν σαφώς τη συμφωνία του Μίνσκ και νομίζω ότι ε, αποτελούν ένα χαστούκι στην διεθνή τάξη. Να ρωτήσω λοιπόν, συνεχίζει στα γαλλικά η κυρία Καλνίεται από τον Γάλλο προλαλήσαντα, εάν θα υποστηρίξει για μια ακόμη φορά την αυτοδιάθεση κάποιων επαρχιών ε, των Βάσκων, ε, των Οξιτανών της Νότιας Γαλλίας εφόσον αναζητηθεί μια τέτοια προσπάθεια αυτονομίας. Νομίζω ότι για σας και για το κόμμα σας κάτι τέτοιο ε, δεν είναι, είναι εκτός πραγματικότητας. Τελειώνοντας λοιπόν θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι που είπε ο Μιχαήλ Χοντορχόφσκι. Ξέρετε ποιος είναι ο Χοντορχόφσκι. Το είπε ρωσικά και θα το πω λίγο, θα το μεταφράσω λίγο ελεύθερα. Εγώ δεν θέλω να μιλήσω για τις προσωπικότητες. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι γιατί όλοι οι παλιοί φασίστες από την Ευρώπη υποστηρίζουν τον Πουτίν. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε κάποια από τα ερωτήματα τα οποία απευθυνόντουσαν σε μένα. Λέει η κυρία Τεσουλουέτα. Το θέμα της εκπροσώπησης των γυναικών. Χαίρομαι που αυτό λαμβάνεται στα σοβαρά. Είναι κάτι το, στο οποίο το Ίδρυμα για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα δίνει μεγάλη σημασία στις εκθέσεις του. Οι γυναίκες με τις οποίες μίλησα στην Ουκρανία απέδωσαν την χαμηλή τους αντιπροσώπευση στον κυρίαρχο χρόνο, κυρίαρχο ρόλο των χρημάτων στην εκλογική διαδικασία και στην πίεση της βίας, που έκανε πολύ πιο δύσκολη τη συμμετοχή τους. Για τους εσωτερικά εκτοπισμένους, το αν υπήρξαν αρκετέ προσπάθειες να καλυφθούν τα άτομα, αυτό, αυτό είναι δύσκολο να το, να το ξέρουμε. Επί βάση όμως της παρατηρητής μας, είδαμε ότι υπήρξε μεγάλη ανισομέρειες. Σε μερικές περιοχές όπως το Χάρκοβο έγιναν σημαντικές προσπάθειες με κάπως βέβαια απογοητευτικά αποτελέσματα. Σε άλλες περιοχές ήταν αντικειμενικά πολύ πιο περιεσμένες οι προσπάθειες αυτές για τη συμμετοχή των νέων. Δεν έχουμε μηχανισμό για να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε αυτή την πτυχή της προεκλογικής διαδικασίας. Θα πρέπει όμως να είμαστε προσεκτικοί πρωτού πούμε ότι οι νέοι εκλογής δεν ε, έλαβαν, χώρα, έλαβαν ε, μέρος στις εκλογές γιατί νομίζω ότι παίξανε μεγάλη, μεγάλο ρόλο στην επιτυχία ενός τουλάχιστον πολιτικού κόμματος. Πιστεύω λοιπόν ότι οι εκλογές ήταν μέσα στα συνηθισμένα σε επίπεδο εκλογών. Τώρα βέβαια υπήρξαν μεγάλες διαφορές σε εσωτερικό επίπεδο. Στα ανατολικά της χώρας ήταν μικρότερη η συμμετοχή. Τώρα, σε σχέση με την επίπτωση της ύπαρξης ένστολων, αυτό είναι κάτι το οποίο το λάβαμε υπόψη μας πολύ προσεκτικά μετά από εκθέσεις και αναφορές για πολλούς ένοπλους και ένστολους και επίσης λόγω του γεγονότος ότι πολλοί επικεφαλής στρατιωτικών τμήματων ήταν υποψήφιοι στις εκλογές σε περιοχές όπως το Λουχάνσκ και το Ντονέτσκ. Αλλά είχαμε μονάχα δύο περιπτώσεις που υπήρξαν, που ανέφεραν παρουσία ένστολων σε εκλογικά τμήματα. Δυστυχώς βέβαια υπήρξαν και περιπτώσεις ένστολων οι οποίοι επηρέασαν ή τουλάχιστον προσπάθησαν να επηρεάσουν την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων Η πρώτη μας λοιπόν ενδιάμεση έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι υπήρξαν περιπτώσεις ε, διακρίσεων και τρομοκρα... τρομοκράτησης ατόμων κυρίως από το προηγούμενο Κομμουνιστικό Κόμμα τα κόμματα όμως της αντιπολίτευσης μας προσέγγισαν πριν και μετά από τις εκλογές, μας είχαν αναφέρει τις ε, ανησυχίες τους και μετά τις εκλογές χρησιμοποιώντας το δικό του σύστημα καταμέτρησης που είναι παράλληλο με το επίσημο θεώρησαν ότι ήταν ε, θετικά τα αποτελέσματα των εκλογών και δεν τα διαμφισβητούν και ευχαριστούν τη διεθνή κοινότητα για την αμερόληπτη παρακολούθηση των εκλογών και τη βοήθειά τους. Για τις ε, εκλογές στο ρωσόφωνο τμήμα υπήρχαν 18 παρατηρητές σε μικτές εθνοτικά ομάδες, αυτή είναι η μεθοδολογία που ακολουθείται και εκεί δεν αναφέρθηκαν προβλήματα, οι περισσότεροι από αυτούς ήταν επεπειραμένοι <clears throat> παρατηρητές και πιστεύω ότι οι αναφορές τους ήταν απόλυτα ευθυγραμμισμένες με τις υπόλοιπες Άκουσα ότι ο Ρώσος Υπουργό Εξωτερικών είπε ότι η Ρωσία αποδέχεται το αποτέλεσμα αυτών των εκλογών. Σε σχέση με το εκλογικό σύστημα και τη μεταρρύθμιση του εκλογικού συστήματος, η ΟΔΙΕ, το Ίδρυμα για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, δεν προωθεί ένα σύστημα σε βάρος των άλλων. Αλλά στην αρχική μας παρέμβαση τονίσαμε ότι παρά τις εκκλήσεις για μεταρρύθμιση του εκλογικού συστήματος και της υποσχέσεις ότι θα γίνει κάτι τέτοιο, το Κοινοβούλιο της Ουκρανίας δεν ενέκρινε αυτήν την ε, μεταρρύθμιση. Εμείς πάντα λαμβάνουμε υπόψη αυτές τις ε, εθνικές προσδοκίες και προσπαθούμε να τις λάβουμε υπόψη όπως και τις προτάσεις της Επιτροπής Βενετίας του Συμβουλίου της Ευρώπης. Και νομίζω τώρα ότι έχω απαντήσει στα σχόλια, τουλάχιστον αυτά θυμάμαι να απευθύνονται σε μένα. Ευχαριστώ. Θα ξεχύσει τον κύριο Νάρτ και θα δώσουμε μετά το λόγο στον κύριο Πλένκοβιτς. Άκουσα με μεγάλη προσοχή τα λόγια του Πρόεδρου Κόουσο και του Γάλλου συναδέλφου, του κύριου Σαφχάουσερ. Και νομίζω ότι προέρχονται από την κοινή λογική. Μπορεί να είναι εναντίον της κυριαρχούσας γνώμης, αλλά περιέχουν κάτι το οποίο είναι ουσιαστικό. Το να θεωρήσουμε το πρόβλημα της Ουκρανίας ένα πρόβλημα σύγκρουσης μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε καμία γνώση της πραγματικότητας. Η Ρωσία προφανώς εμπλέκεται στο θέμα αυτό. Αλλά δεν μιλάμε για ένα εξωτερικό φορέα και ένα εσωτερικό φορέα γιατί ένας από τους εσωτερικούς παράγοντες στην Ουκρανία που υποστηρίζεται από ένα τμήμα του πληθυσμού είναι η Ρωσία. Νομίζω ότι με μια τέτοια μανιχαϊκή αντιμετώπιση δεν πρόκειται να καταλήξουμε πουθενά. Υπάρχει κάτι το οποίο είναι αδιαμφισβήτητο, ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε την ενότητα και την εδαφική ακαιρεότητα της ε, Ουκρανίας. Αυτό θα πρέπει να είναι ο οδηγό μας και για την Ουκρανία και στη Μολδαβία και στη Γεωργία όταν αντιμετωπίζουμε σοβαρά εσωτερικά προβλήματα. Είναι μια πραγματικότητα που δεν είναι απλή. Έχουμε τον κατακαιρματισμό της πρώην Σοβιετικής Αυτοκρατορίας σε διοικητικά όρια τα οποία είναι εθνικά όρια και τα οποία πρέπει να τα διατηρήσουμε ως έχουν, αλλιώς θα διαλυθεί και η συμφωνία του Ελσίνκη και θα καταρρεύσει η Ευρώπη και σας υπενθυμίζω την περίπτωση του Κωσυφοπεδίου που ήταν η περίπτωση αυτή που άνοιξε το κουτί της Πανδώρας. Θα πρέπει να υπάρξει μια λύση λοιπόν ουκρανική η οποία να βασίζεται στην ενότητα και την εδαφική ακαιρεότητα της Ουκρανίας. Αν το μόνο όμως το οποίο έχουμε στο μυαλό μας είναι ένας κακόβουλος εξωτερικός εισβολέας, τότε θα δουλεύουμε με καρικατούρες και δεν θα καταλήξουμε ποτέ σε μια πραγματική λύση. Πρέπει λοιπόν να έχουμε και την πραγματικότητα υπόψη μας. Υπάρχουν ορισμένοι που λένε ότι αν η πραγματικότητα διαψεύδει τις ιδέες μας, τότε τόσο χειρότερο για την πραγματικότητα δεν σύμφωνο με αυτό. Κύριο Σαφχά. για αν θέλετε να λάβει το λόγο. Ναι κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Φυσικά και πάντα εγώ είμαι υπέρ της ενότητας του κράτους και γι' αυτό άκουσα προσεκτικά αυτά που είπε η συνάδελφος. Αλλά δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη αν δεν υπάρξει πράγματι ενότητα της Ουκρανίας. Η ενότητα αυτή όμως ε, καθίσταται όλο και πλέον δύσκολη. Έχουμε μια νέα πραγματικότητα μπροστά. Η χώρα αυτή έχει το αίσθημα ότι υπέστη μια επίθεση και σύν της άλλης ε, ο λαός βλέπει ότι ε, κατά κάποιο τρόπο αγνοείται μερικές φορές από την πολιτική εξουσία και αυτό οδηγεί σε κάτι το οποίο δεν επιθυμούμε, αλλά το οποίο τελικά θα είναι αυτό που ονομάζουμε απόσχηση. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο συνέβη και στο κοσυφοπαίδιο. Η πολιτική των δύο στάνταρ, των δύο επιπέδων ε, είναι καταδικαστέα. Εγώ είμαι υπέρ της ενότητας όλων αυτών των χωρών αλλά να πω ότι οι περιοχές αυτές ε, της Ανατολικής Ευρώπης, αν κοιτάξουμε την μακρά ιστορία, ανήκαν στην ε, Ρωσία. Και ο Στάλιν είναι αυτός ο οποίος τροποποίησε τα σύνορα. Εγώ δεν είμαι υπέρ του να θεωρήσουμε ότι τα σύνορα του Στάλιν είναι αυτά τα οποία θα πρέπει να επικρατήσουν. Πρέπει να ξεκινήσει επιτέλους ένας ουσιαστικός διάλογος και ο διάλογος αυτός δεν μπορεί να υπάρξει παρά μόνον αν αναγνωρίσουμε μια κάποια νομιμότητα και στις εκλογές της Ανατολικής Ουκρανίας αλλά να υπάρξει διάλογος. Αυτό απαιτεί η ε, συγκεκριμένη περίπτωση και η ειρηνευτική προσπάθεια. Προτού δώσω το λόγο στην κυρία Ντόρις Πακ, λέει ο πρόεδρος, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Πλέγκοβιτς. If Doris would like to speak first, I have no Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι ήταν μια πάρα πολύ λεπτομερής και χρήσιμη συζήτηση και των γεγονότων που έλαβαν χώρα και χθες πρέπει να υπογραμμίσουμε το πάρα πολύ σημαντικό έργο της Εκλογικής Επιτροπής, της ε, Εθνικής Εκλογικής Επιτροπής στην ε, Ουκρανία, που έδωσε δυνατότητα σε αυτούς οι οποίοι προέρχονται από τις λεγόμενες κατεχόμενες περιοχές του Λουχάνς και του Ντονέτσκ να μπορέσουν να λάβουν μέρος στις εκλογές. Θέλω να τονίσω επίσης ότι πέραν των συναντήσεων μας με τους πολιτικούς συνομιλητές μας είχαμε συζήτηση και με τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών ήταν πάρα πολύ σημαντική αυτή η συζήτηση και από την αρχή της διαδικασίας του Ευρωμαϊντάν πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να υποστηρίξει αυτές τις διαδικασίες. Ήταν επίσης σαφές ότι το θέμα της εδαφικής ακαιρεότητας είναι απαράγραπτο. Αυτό είναι κάτι που η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα πρέπει ποτέ να δεχτούν ως τετελεσμένο γεγονός. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να είναι σαφείς οι μας. Γι' αυτό Θέλω να τονίσω ότι είναι απαραίτητο να εξασφαλίσουμε την ε, ταχεία συγκρότηση της νέας Βέρχοβαράντα του Κοινοβουλίου της Ουκρανίας και της κυβέρνησης, γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να υποστηρίξουμε αυτές τις ευρωπαϊκόστροφες μεταρρυθμίσεις που είναι απαραίτητες για την Ουκρανία και να διατηρήσουμε το πνεύμα ειρήνης που ήταν αυτό το οποίο ήταν το βασικό νόημα των εκλογών. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πλέγκοβιτς για την ε, σύνοψή σας αν μπορώ και εγώ να κάνω κάποια σχόλια. Εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως και η Ουκρανική Ράντα, έχουμε κυρώσει τη Συμφωνία Σύνδεσης, που προέβλεπε και τις εκλογές της 25ης Οκτωβρίου, ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης νομιμοποίηση του Κοινοβουλίου και της κυβέρνησης της Ουκρανίας. Έχουμε λοιπόν να, το καθήκον να εξασφαλίσουμε την εφαρμογή αυτών των συμφωνιών. Ήταν μια δύσκολη κατάσταση διότι ξεκινήσαμε σε συνθήκες ε, ένοπλης αντιπαράθεσης αλλά πιστεύω ότι η γενική κρίση των ε, παρατηρητών είναι ότι ήταν πολύ καλές οι συνθήκες των εκλογών. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι θα πρέπει να δεχτούμε πλήρη την νομιμοποίηση της κυβέρνησης της Ουκρανίας μετά από αυτές τις εκλογές. Πιστεύω επίσης ότι πρέπει να συνεχιστούν και οι συζητήσεις με την Ρωσία επί τη βάση της συμφωνίας του Μίνσκ. Οι χθεσινές τώρα εκλογές ήταν μια παραβίαση συμφωνίας του Μίνσκ. Αυτό για μένα είναι αναμφίβολο. Και επομένως είναι μια η παναχώρηση για τη διαδικασία του Μίνσκ. Θα πρέπει λοιπόν να επιμείνουμε στο ότι δεν έχουμε μόνο ένα εσωτερικό πρόβλημα στην Ουκρανία, αλλά έχουμε τα γεγονότα τα οποία έχουν γίνει στην Κρυμαία και την Ανατολική Ουκρανία, που είναι γεγονότα τα οποία έχουν προκληθεί από μια εξωτερική επέμβαση. Πρέπει λοιπόν να λαμβάνουμε υπόψη ότι πρέπει να τηρούνται τα πρότυπα σε όλες τις εκλογές. Δεν μπορούμε να έχουμε λοιπόν μια διαφορετική αντιμετώπιση σε, για τις εκλογικές διαδικασίες. Νομίζω ότι γνωρίζουν ορισμένοι κάποια συστήματα περισσότερο από άλλα. Δεν πρέπει να παρασύρεται κανείς από αυτά τα οποία του είναι προσφυλή. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε απόλυτα ομοιόμορφα τις ε, διαδικασίες εκλογών. Παρά την ε, ε, πρόταση του πρόεδρου Ποροσέγκο να γίνουν και στις περιοχές αυτές εκλογές επί τη βάση του Ουκρανικού δικαίου. Αυτό είναι φανερό ότι δεν έγινε δεκτό από τη, τους ε, ασκούντες στην εξουσία στις ανατολικές επαρχίες και αυτό δημιουργεί τις δυσκολίες που έχουμε ενώπιόν μας. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να έχουμε μια συμφωνία με τη Ρωσία, θα πρέπει όμως να είναι σαφές ότι το διεθνές δίκαιο δεν παραβιάστηκε από την Ουκρανία αλλά από την Ρωσία και αυτό θα πρέπει να είναι και η βάση με την οποία θα προχωρήσουμε και επί τη βάση της ε, συμφωνίας του Μίνσκ η οποία πρέπει και αυτή να τηρηθεί και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τη συνέπεια της συμφωνίας του Μίνσκ για την Ανατολική Ουκρανία. Και εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είμαστε αποφασισμένοι για την τήρηση της διαδικασίας του Μίνσκ. Θέλω να ευχαριστήσω τους τον εισηγητή και τους ε, άλλους ομιλητές και μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο της τη διάταξης που είναι το θέμα του κοσφοπεδίου. Ξέρουμε ότι υπάρχουν και από το Κόσοβο αναφορές Υπάρχουν,